Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Ισπανίδα Υπουργό Γεωργίας και να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση. Ε, για τα ζωοτεχνικά θέματα. Έχουμε ένα ντοσιέ με δύο σημεία. Καταρχήν, το κανονισμό για τον οποίο η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Νταντέ, τον οποίο θα αρχίσουν ε, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Αφορά το εμπόριο ε, ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Και το δεύτερο αφορά την ε, απλουστευμένη διαδικασία θα έλεγα να αναβάλουμε για την επόμενη μας συνεδρίαση την ψηφοφορία για την απλουστευμένη διαδικασία. Και περνάμε τώρα στο κύριο θέμα που σας είπα της σημερινής ημερήσιας διάταξης που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την Ισπανίδα Υπουργό Γεωργίας, την κυρία Ιζαμπέλ Γκαρσία Τεχερίνα. Με θέμα της ε, εμπειρίας της Ισπανίας, σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του νομο, του, της νομοθεσίας για τον έλεγχο της επιστηστικής αλυσίδας, της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό και για την καλοσύνη που είχε να έρθει στη συνεδρίαση και να μας παρουσιάσει τις εμπειρίες της πατρίδας της, της Ισπανίας, ε, μετά την εφαρμογή του Ισπανικού νόμου για την επισητιστική αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ πριν από μία διετία. Είναι επίκαιρο το θέμα γιατί και εμείς ασχολούμαστε με το θέμα της καταπολέμησης των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην επισητιστική αλυσίδα και διαρωτόμαστε κατά πόσο χρειάζεται και κοινοτική νομοθεσία για το θέμα αυτό. Γι' αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε την ε, παρουσίαση της ισπανικής εμπειρίας στα θέματα αυτά. Είναι ιδιαίτερα επίμαχο το θέμα και προτείνονται διαφορετικές λύσεις. Μάλιστα έχουμε προχωρήσει με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο μέχρι στιγμής στις συζητήσεις. Γι' αυτό και με μεγάλη ικανοποίηση θα ακούσουμε την παρουσίαση της ισπανικής εμπειρίας στα θέματα αυτά. Η Ισπανία άλλωστε είναι η χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο στα θέματα αυτά, είναι η πιο πρωτοπόρα και θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε θερμά και να εκφράσω και πάλι τη χαρά μας γιατί με τέτοια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Υπουργών και Ευρωβουλευτών βελτιώνονται οι σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Γιατί, όπως σας είπα, παράλληλα έχουμε και εμείς ε, αντίστοιχες ε, συζητήσεις. Αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ΙΜΚΟ και εμείς ε, θα συντάξουμε γνωμοδότηση. Η κυρία Μαγκίνες έχει αναλάβει το θέμα αυτό. Φαντάζομαι θα λάβει το λόγο αργότερα στην ανταλλαγή απόψεων, αλλά ήρθε η ώρα να σας δώσουμε το λόγο κύριε Υπουργέ για να μας κάνετε την παρουσίασή σας που θα την ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. να μας περιγράψετε τις εμπειρίες της Ισπανίας από το θέμα του νόμου για τον έλεγχο της επιστημιστικής αλυσίδας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην συνεδρίασή σας και στην Επιτροπή σας και θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν και που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για μία ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα προβλήματα που δημιουργούν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Και φυσικά, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια βήματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υιοθετήσουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων από τις αθέμητες πρακτικές. Από το Υπουργείο Γεωργίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ισπανίας παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή τι διάφορε εργασίε και τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ε, και μάλιστα πρόκειται για έγγραφα όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Κοινωνική και οικονομική επιτροπή. Στα έγγραφα αυτά και επανειλημμένως επισημάνθηκε η σημασία του προβλήματος και οι αρνητικές συνέπειες αυτών των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Δεδομένου του περιεχομένου των εγγράφων αυτών, αλλά και των απόψεων των διαφόρων φορέων της επιστηστικής αλυσίδας και των αρμόδιων εθνικών αρχών για το θέμα αυτό, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων ως προς τη διάγνωση της κατάστασης και την σοβαρότητα του προβλήματος. Επιτρέψτε μου τώρα να απαριθμίσω ορισμένα σημεία που κατά τη γνώμη μου μας ε, επιτρέπουν να κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές εμφανίζονται κυρίως ως συνέπεια της διαφοράς ε, που υπάρχει στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των διαφόρων κρίκων της επιστημιστικής αλυσίδας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως ε, οι αγρότες ε, παραγωγή και η κτηνοτρόφη παραγωγή εκτίθενται ιδιαίτερα, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και αυτό παρεμποδίζει την μελλοντική τους βιωσιμότητα και περιορίζει τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που γίνονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση και ολοκλήρωση, ιδιαίτερα στον τομέα της διανομής, αυξάνουν τις διαφορές αυτές στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των διαφόρων φορέων αυτής της αλυσίδας. Κάτι που αυξάνει την τροτότητα των παραγωγών, αλλά και των μεταποιητών, σε μικρότερο βαθμό όμως. Υπάρχει ομοφωνία ως προς, την, τον αρνητικό αντικτύπο των αθέμητων πρακτικών στις επενδύσεις και την καινοτομία εκ μέρους των επιχειρήσεων, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέλος, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, συνιστούν ένα εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της ευρωένιας αγοράς και στρεβλώνουν τους μηχανισμούς της αγοράς. Οπότε, εν κατάστασης, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρότριναν τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν λύσεις προκειμένου να προστατεύσουν τους ε, μικροεπιχειρηματίες και κυρίως ε, τους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Οπότε οι αρμόδιες αρχές προβληματίζονται για το ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Διαπιστώνουμε πάντως ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα των εμπορικών πρακτικών, των αθέμητων εμπορικών πρακτικών μεταξύ των διαφορών χωρών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πώς η Ισπανία αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό και ποιο είναι το μοντέλο που εφαρμόζουμε και που αρχίζει ήδη να αποφέρει καρπούς. Ε, η... Έχουμε αναλάβει την εξουσία εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια με την κυβέρνηση του Λαϊκού και δείξαμε ιδιαίτερη ευαισθησία στην ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη στην οποία βρίσκονται οι μικροί παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι και διαπιστώσαμε την ανισορροπία που υπάρχει στην επιστηστική αλυσίδα εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των τιμών ή εξαιτία εφαρμογή ε, αθέμητων εμπορικών πρακτικών ε, εκ μέρου κάποιων φορέων τη επιστημιστική αλυσίδα. Γι' αυτό και αναλάβαμε τη δέσμευση να υποβάλουμε προτάσεις για μια πιο βιώσιμη, πιο ισορροπημένη επιστημιστική αλυσίδα και αλυσίδα αξιών και να προστατεύσουμε τους ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένοι και μέχρι στιγμής ήταν υποχρεωμένοι να παραδίδουν την παραγωγή τους χωρίς συμβάσεις, ε, χωρίς καθορισμό τιμής και χωρίς να γνωρίζουν πότε θα εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται. Έτσι λοιπόν εργαστήκαμε άοκνα για να εκπονήσουμε ένα νομοσχέδιο με ζητούμενο τη συνένεση και διαβούλευση με όλους τους κρίκους της επιστηστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και φροντίσαμε να έχουμε επαφές με όσες οργανώσεις ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας ε, φροντίζοντας να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα είχαν ε, ευρεία συνένεση. Αποτέλεσμα ήταν το, ο νόμος 12 το 2013 για τα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας της επιστημιστικής αλυσίδας που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης στις 2 Αυγούστου του 2013. Στόχος είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και αντιγωνιστικότητα του αγροεπιστημιστικού τομέα, να μειωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων κρίκων της αλυσίδα ε, αξιών και να διαμορφωθεί ένα δίκαιο πλαίσιο που θα επηρεάζει ε, και θα ωφελεί όχι μόνο τους φορείς της επιστηστικής αλυσίδας αλλά και τους καταναλωτές. Η εφαρμογή ε, και η θέση ισχύ του νόμου βελτίωσε τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κρίκων της επιστήστικης αλυσίδας και μάλιστα η βελτίωση αυτή ήταν άνευ στην Ισπανία ε, νομίζω ότι είναι ανευπροηγουμένου και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος 12 του 2013 θέσπισε ένα νέο νομικό πλαίσιο, πιο δίκαιο και ισορροπημένο, το οποίο ισχύει για τις εμπορικές σχέσεις όλων των φορέων της ε, επιστηστικής αλυσίδας, ξεκινώντας από την παραγωγή και καταλήγοντας στην διανομή που φέρει τα τρόφιμα στη διάθεση των πολιτών. Έχουμε ένα μεικτό μοντέλο στο νόμο, με τη συνύπαρξη ενός δημοσίου συστήματος που ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και ενός ιδιωτικού συστήματος αυτορύθμισης που θεσπίζει το πλαίσιο για πιο ποιοτικέ εμπορικές σχέσει που συμπληρώνονται από ένα σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας ώστε να εντοπίζουμε τα προβλήματα όταν ανακύπτουν και να διαπιστώνουμε την, τις εξελίξεις ό,τι αφορά την ποιότητα των εμπορικών σχέσεων. Θα ήθελα τώρα με κάποιες λεπτομέρειες να σας παρουσιάσω τα πέντε στοιχεία αυτού του νέου μοντέλου του νέου νόμου για την επισητιστική αλυσίδα. Καταρχήν, στα πλαίσια του δημοσίου συστήματος ρύθμισης, θα ήθελα να πω ότι από την αρχή κρίναμε ότι για να είμαστε αποτελεσματικοί στη βελτίωση της επιστημιστικής αλυσίδα έπρεπε να ρυθμίσουμε τις ε, βασικές εμπορικές πρακτικές και να ορίσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Έτσι, ο νόμος ε, προβλέπει κάποιες πρακτικές που θεωρούνται υποχρεωτικές, όπως είναι η ε, υποχρεωτικός χαρακτήρα σύναψης σύμβασης για τις εμπορικές σχέσεις οι συμβάσει αγοραπολισία θα πρέπει να επισημοποιούνται και γραπτώ σε περίπτωση που ένα φορέα είναι αγρότη παραγωγό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση αδυναμίας απέναντι στο συμβαλόμενο μέρος. Χάρη στις ρυθμίσεις αυτές ε, είχαμε σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές αλλαγές ε, που κατά παράδοση ταλάνιζαν τους αγρότες γιατί ε, δεν πρόβλεπαν καθορισμό τιμών ή δεν προέβλεπαν εχέγγυα για την ε, ανάκτηση ε, του τιμήματος. Οπότε τώρα με τις νέες ρυθμίσεις οι αγρότες θα γνωρίζουν τι τιμή θα εισπράξουν για το προϊόν τους και πότε. Προβλέπονται και κάποιες ε, προϋποθέσεις ε, για την εφαρμογή κάποιων πρακτικών, όπως είναι οι πληστηριασμοί μέσω διαδικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια στις πρακτικές αυτές. Επίσης απαγορεύονται κάποιες καταχρηστικές πρακτικές, όπως η μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων, για παράδειγμα, η, η απέτηση εμπορικών δασμών που δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή, η απέτηση να παρασχεθούν εμπορικά ευαίσθητες πρωτο... Ε, πληροφορίες, η εφαρμογή πρακτικών που αντιβαίνουν στον ε, υγιή ανταγωνισμό, η διαχείριση σημάτων, η εκμετάλλευση υπέρ κάποιων φορέων ε, ξένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ορισμό των αθέμητων πρακτικών, γι' αυτό και ήταν απαραίτητο να προβλέψουμε εκτός από τον ορισμό και ένα σύστημα κυρώσεων καθώς και ένα σύστημα ελέγχου. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Οι δέσμοι των κυρώσεων που ισχύουν, μερικές φορές είναι πολύ αυστηρές, φτάνουν και μέχρι το 1 εκατομμύριο ευρώ και μάλιστα ε, ιδρύσαμε και έναν οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εφαρμογής αυτών των πρακτικών και της ε, εφαρμογής των κυρώσεων. Γι' αυτό και έχουμε τον οργανισμό για τις πληροφορίες και τον έλεγχο σε θέματα τροφίμων τον οργανισμό ΑΙΚΑ. Δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν από τον παράγοντα φόβο, γι' αυτό και πολύ δύσκολα οι αγρότες ε, κάνουν καταγγελίες για καταχρηστικές συμπεριφορές, ο νόμος προβλέπει ότι τέτοιες καταγγελίες ε, εκτός από τους άμεσα θυγόμενους μπορούν να υποβάλλονται και από ενώσεις παραγωγών και μάλιστα ακόμη και ανώνυμα. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα να ξεκινούν αυτεπάγγελτα από τον Οργανισμό Πληροφορίας και Ελέγχου μίας ε, ε, έρευνας για να ανοιχνευτεί μια τέτοια καταχρηστική συμπεριφορά. Δεν θέλαμε λόγω προβλημάτων επικοινωνίας με τις αρχές ε, να μείνουν χωρίς συνέχεια τέτοιες καταχρηστικές συμπεριφορές. Επίσης έγινε μια τυποποίηση των κυρώσεων με προοδευτικό τρόπο. Σε περίπτωση ε, κατεξακολούθηση εφαρμογής ε, καταχρηστικών συμπεριφορών οι κυρώσεις γίνονται ακόμη πιο αυστηρές. Στην αρχή θέλαμε να, κάνουμε, να δώσουμε προειδοποίησεις με αποτρεπτικό χαρακτήρα κάποιων ελαφρών σχετικά επικών κυρώσεων, οι οποίες γίνονται όλο και πιο αυστηρές στο μέτρο που επαναλαμβάνεται η εφαρμογή των καταχρηστικών συμπεριφορών και επαναλαμβάνω η πιο αυστηρή κύρωση είναι η επιβολή χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου ευρώ σε περίπτωση που έχουμε καταξακολούθηση τέτοια ε, συμπεριφορά. Προβλέπεται μάλιστα μια μέγιστη προθεσμία έξι μηνών για τη διεκπαιρέωση τέτοιων υποθέσεων, ώστε από την υποβολή της, καταγγελίας σχετικά σύντομα έχουμε την ε, διεκπαιρέωση της ε, υπόθεσης. Και μάλιστα, επειδή η δημόσια διοίκηση αναλαμβάνει τη διαχείριση και την έρευνα τέτοιων περιπτώσεων, η εφαρμογή ε, αυτών των μέτρων του νόμου γίνονται χωρίς κόστος για τον καταγγέλλοντα. Και οι ενδιαφερόμενοι και η δημόσια διοίκηση έχουν ε, αναποθέσει όλες τις ελπίδες στο σύστημα αυτό. Και μάλιστα και η παραγωγή και οι διάφοροι φορείς επιστημιστικής αλυσίδας βρίσκουν σε αυτόν τον οργανισμό ελέγχου και πληροφοριών το μεγαλύτερο θεματοφύλακα της νομιμότητας. Ήταν πολύ επιτυχημένη η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Για παράδειγμα, ε, λύθηκαν τα προβλήματα στον τομέα απορροκυπευτικών εξαιτία του ρωσικού βέτο. Γιατί χάρη στην εφαρμογή ε, αυτού του ελέγχου μπορέσαμε να απαλείψουμε κάποιες κακές ε, εμπορικές πρακτικές που επιβάρυναν τους παραγωγούς και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση με το ρωσικό εμπάργο που έπληξε ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, τον τομέα των οπορεκυπευτικών στην Ισπανία. Σε ό,τι αφορά τον γαλακτοκομικό τομέα, ο νόμος αυτός συμπλήρωσε την κοινοτική νομοθεσία για τις ενοχικές σχέσεις που προβλέπει ο κανονισμός της κοινή οργάνωσης αγοράς ε, ε, προϊόντων. Η Ισπανική νομοθεσία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ε, αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία και έτσι ε, συγκεντρώσαμε πολύ χρήσιμε πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις σε ένα πολύ σημαντικό τομέα όπως είναι αυτός των γαλακτοκομικών προϊόντων. Διαπιστώσαμε ότι θα έπρεπε και εδώ να έχουμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς κυρώσεων που θα ισχύουν στις ε, συμβάσεις του γαλακτοπαραγωγικού τομέα που είναι ένα τμήμα των συμβάσεων της επιστημιστικής αλυσίδας. Έτσι ενισχύσαμε την εφαρμογή των συμβάσεων και την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων. Και όλα αυτά υπέρ της, ε, του πιο τροτού κρίκου της αλυσίδας που είναι η κτηνοτρόφη. Έτσι χάρη στον οργανισμό ΆΙΚΑ και χάρη στην νομοθεσία αυτή ο Οργανισμός ε, Ελέγχου και Πληροφοριών είναι από το 2015 ο αρμόδιος για το συντονισμό των ελέγχων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των, υποχρεώσεων, ε, των ενοχικών υποχρεώσεων στον γαλακτοκομικό τομέα και να εφαρμοστούν ε, στο έπακρο οι αυτές. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που έχουμε ε, συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, διαπιστώνουμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο που λειτουργεί αυτή η ΑΕΚΑ, ο Οργανισμός δηλαδή Ελέγχου και Ενημέρωσης, Έχουμε ελέγξει αυτεπάγγελτα 663 ε, επιχειρήσεις και 3.000 εμπορικές συναλλαγές. 91 καταγγελίες έχουμε λάβει για μη συμμόρφωση με το νόμο, κυρίως ε, καταγγελίες που έχουν γίνει από ενώσεις παραγωγών ε, και μετά τις καταγγελίες αυτές ε, ξεκίνησαν 141 υποθέσεις επιβολής κυρώσεων. Το τρίτο στοιχείο του νόμου μας προβλέπει ένα σύστημα αυτορύθμισης που αυξάνει σημαντικά το πεδίο προστασίας πέραν των υποχρεωτικών διατάξεων. Αυτό το επιτυχάνουμε χάρη σε ένα κώδικα καλών εμπορικών πρακτικών στις συμβάσεις ε, της επιστηστικής αλυσίδας. Έτσι, με προαιρετικό και οικιοθελή τρόπο, διευρύνουμε τις υποχρεώσεις των διαφόρων φορέων της αλυσίδας, πέραν αυτών που προβλέπονται από τον νόμο, ώστε να βελτιώσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης ε, μεταξύ των εμπορικών τελεστών. Καλούμε ε, τις επιχειρήσεις της παραγωγής, ε, της βιομηχανίας, ε, της διανομής και της ενώσης τους να προσχωρήσουν σε αυτόν τον κώδικο. Και ναι μεν είναι προαιρετική η προσχώρηση σε αυτόν τον κώδικα καλών πρακτικών, δίνονται κίνητρα για να ενισχυθεί αυτή η προσχώρηση. Και μετά από διετής προσπάθειες καταλήξαμε πρόσφατα σε αυτόν τον κώδικα καλών πρακτικών με τις ενώσεις ε, γεωργών, τους συνεταιρισμούς, του αγροεπιστιστικό κλάδο και τον κλάδο των διανομέων. Πρόκειται για ένα κείμενο που απαρτίζεται από 50 άρθρα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των υποχρεώσεων τις οποίες προαιρετικά αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις τους. Το τέταρτο στοιχείο της Ισπανικής νομοθεσίας αφορά ένα ισχυρό σύστημα επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνεται στον κώδικα βέλτιστων πρακτικών και που δίνει άμεση απάντηση και μάλιστα με σχετικά χαμηλό κόστος και με εχέγγυο αμεροληψίες στις πιθανές διαφορές που ίσως προκύψουν από τη μη συμμόρφωση ή την αθέτηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των συμβαλωμένων. Η θέση ισχύ του συστήματος επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται στον κώδικα αυτό δίνει νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εμπορικών τελεστών, όπως θα συμβεί και με την ε, ανάληψη των ε, καθηκόντων από τον νέο μεσολαβητή που θα μπορεί να επεμβαίνει μετά από έτσι των ε, συμβαλωμένων μερών ή των ενώσεων για να καθοριστούν οι τιμές μεταπημένων προϊόντων. Επίσης προβλέπεται στον κώδικα και το αξίωμα του συνηγόρου, του πελάτη και του προμηθευτή, που θα είναι το πρώτο επίπεδο επίλυσης των διαφορών. Επιπλέον, ο κώδικας προβλέπει την υποχρέωση των ε, διαφόρων φορέων να επιλύουν τα προβλήματα και τις διαφορές τους ε, καλή την πίστη και με χαμηλό κόστος με βάση κάποια μοντέλα διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Κατά την εκπόνηση του σχετικού νομοσχεδίου μας ε, απασχόλησε η βιωσιμότητα αυτού του νόμου και η διάρκεια του μέσα στον χρόνο. Γι' αυτό και το σύστημα που προβλέπουμε συμπληρώνεται από ένα σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας ολόκληρου του αγοροπιστικού τομέα έχουμε το παρατηρητήριο της επιστημιστικής αλυσίδας που αποτελεί και το πέμπτο στοιχείο του νόμου αυτού. Και χάρη στο έργο του σχετικού παρατηρητηρίου μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου και να εντοπίσουμε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Συγκεντρώνουμε έτσι πληροφορίες ε, για τη δημιουργία των προβλημάτων, την εμφάνιση κάποιων νέων και τις εξελίξεις στην ποιότητα των εμπορικών σχέσεων. Γενικά με το παρατηρητήριο αυτό της επισητιστικής αλυσίδας ε, καταφέραμε να εντοπίσουμε κάποιους τομείς στους οποίους ε, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση επικαιροποιώντας συνεχώς τον νόμο μας. Βέβαια, ο νόμος αυτός είναι σχετικά καινούριος, οπότε δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ήδη γινόμαστε μάρτυρες σημαντικών αλλαγών που πριν από μία τετραετία θα μας φαινόταν αδιανόητες. Δεδομένου όμως ότι αλλάζουμε πρακτικές και συνήθειες πολύ βαθιά ριζωμένες ε, στην ισπανική Ανατροπία, θα χρειαστούν ε, πολλές προσπάθειες, κόπος και χρόνος, αλλά είμαι πεπισμένη ότι βαίνουμε στο σωστό δρόμο και θα επιτύχουμε τους στόχους μας πέραν των προτεραιμάτων του νόμου που συγκεντρώνει σε ε, ένα νομοθέτημα όλα αυτά τα στοιχεία, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του νόμου και ίσως και το κλειδί της επιτυχίας του έγκυται στο γεγονός ότι είναι ένας νόμος για όλους, για όλους τους εμπορικούς τελεστές και όλοι συμμετείχαν στην εκπόνηση του νόμου. Πρόκειται για έναν νόμο που δεν αποκλεί κανέναν, που εφαρμόζει ισορροπημένη ε, αντιμετώπιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των εμπορικών τελεστών, άσχετα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Χάρη στο όνομα αυτό προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε ε, εκ μέρους όλων των κρίκων της αλυσίδας ότι θα πρέπει να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της επιστηστικής αλυσίδας και να θεωρούνται σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι στη διαδικασία της, του εφοδιασμού των τροφίμων. Θα συμφωνείτε ότι ακριβώς επειδή οι διάφορες αλυσίδες αξιών προχωρούν με το ρυθμό του ασθενέστερου κρίκου τους, για να έχουμε ισορροπημένη ισορροπία αυτών των αλυσίδων θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των κρίκων της αλυσίδας ταυτόχρονα. Θα ήθελα εγκατακλείδη να σας αναφέρω τους στόχους που έχουμε επιτύχει χάρη στη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού και που ευελπιστούμε ότι θα επεκταθούν και στο μέλλον, στο μέτρο που αξιοποιούμε όλε τι δυνατότητε τη νομοθεσία. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισορροπία των εμπορικών πρακτικών και να αποφύγουμε τι ε, πρακτικέ αθέμη του ανταγωνισμού, προκειμένου να μην ε, ευνοείται ένας μόνο εμπορικός τελεστής. Θέλουμε μια πιο ισορροπημένη κατανομή της αξίας ε, στις διάφορους κρίκους της αλυσίδας. Ε, θέλουμε να βελτιώσουμε την διαπραγματευτική ικανότητα των παραγωγών, γιατί μετά τη διαφύλαξη των ε, δικαιωμάτων τους ενισχύεται η θέση τους στην επιστημιστική αλυσίδα και βρίσκονται σε καλύτερες συνθήκες για να έχουν καλύτερη διαπραγμάτευση και μεγαλύτερο κέρδο. Θέλουμε επίση πιο εύρυθμη λειτουργία τη αγορά με ενίσχυση τη καινοτομία και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι ο νόμος μας είναι πολύ καλός και θα συμβάλλει σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του αγορεπιστικού τομέα στην Ισπανία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας εκφράσω την προθυμία μου για τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, διαβεβαίωσα και τον Επίτροπο Χόγκαν για την ε, προθυμία μου να συνεργαστώ μαζί του, γιατί θεωρώ ότι όλες αυτές οι εμπειρίες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς που θα ε, ευνοεί τις ε, καινοτόμες ε, προσπάθειες των επιχειρήσεων, γιατί κάτι τέτοιο θα επηρεάσει θετικά το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φέρει σε καλύτερη θέση τις παραγωγές, την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξωτερικές αγορές. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες και πολύ χειροπιαστές. Διαπιστώσαμε ότι σας χαρακτηρίζει και θάρρος και αποφασιστικότητα. Βέβαια, είναι διαφορετικές οι αντιδράσεις και των κρατών και των διαφόρων ε, οργάνων. Μερικοί μιλούν ακόμη και για παρεμπόδιση της ενιαίας αγοράς. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εμπειρίες της Ισπανίας και πολύ καλό παράδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση και για υπόλοιπε χώρες. Ως συνήθως θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές. 14 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι. Δεν θα ήθελα να σας διακόπτω απότομα. Θα σηκώνω διακριτικά το σφυράκι μου για να ξέρετε ότι έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Ο κύριος Αλμπερντές έχει πρώτα το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την ε, Υπουργό Γεωργίας ε, Ιζαμπέλ Γκαρθία Τεχερίνα. Χαίρομαι που ήρθατε και ομολογώ ότι το πρόγραμμά σας ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα. Η κυρία Μαγκίνες επεξεργάζεται το θέμα για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και παρακολούθησε πολύ προσεκτικά επίσης αυτά που μας είπατε, γιατί πολλά από αυτά θα επηρεάσουν και τις δικές μας εργασίες. Είναι ενδιαφέρον πόσες εθνικές δυνατότητες υπάρχουν. Εγώ κάλεσα και το δικό μας Υπουργό επανειλημμένα στη Γερμανία να ακολουθήσει παρόμοια ε, διαδικασία και άλλη μια φορά θα τον ενθαρρύνω ώστε να αξιοποιήσει τις εθνικές δυνατότητες. Και πολύ σωστά είπατε ότι η αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος που συνήθως είναι η παραγωγή. Ε, μια ε, ένωση γαλακτοπαραγωγών μπορεί να έχει 1900 μέλη που παράγουν και πολλούν και πάλι ε, απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες ε, δεν έχουμε την ίδια ισχύ. Θα ήθελα να ρωτήσω, οι εμπορικές αλυσίδες ε, τι ρόλο παίζουν ή τι ρόλο έπαιξαν, συνεργάστηκαν πρόθυμα ή εξαναγκάστηκαν. Ε, επίσης οι προθεσμίες πληρωμής θα πρέπει να μειωθούν αναφέρατε και αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσατε να μας πείτε πόσο μεγάλες είναι οι προθεσμίες πληρωμής στον οποροκυπευτικό τομέα για παράδειγμα. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον για μας. Επίσης μιλήσατε για ένα μοντέλο κυρώσεων που το βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση γιατί αν δεν υπάρχουν κυρώσεις και το όλο σύστημα λειτουργεί εθελοντικά δεν θα είναι τόσο αποδοτικό. Μιλήσατε επίσης για έλεγχο της επιτυχίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Είμαι πρόθυμος και εύχομαι και θα ήθελα το μοντέλο σας να το πάρουμε και γραπτά γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τις περαιτέρω εργασίες μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια των προσπαθειών σας και ελπίζω και από την πλευρά του ΕΛΚ να έχουμε ένα παρόμοιο σύστημα για να λειτουργήσουμε σε παρόμοια βάση. Ευχαριστώ κύριε Δεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητή Ζαμπέλ, καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα αυτή παρέμβαση στην οποία αναφέρθηκε στην ισπανική εμπειρία σε μια πραγματικά ιδιάζουσα στιγμή για μας μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα θα ψηφίσουμε το, την έκθεση της κυρίας Μεγίνες για τις αθέμητες πρακτικές. Συνεπώς θα έλεγα ότι είναι θαυμαστία αυτή η σύμπτωση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που το Κοινοβούλιο μιλάει για τις αδέμητες πρακτικές στην ε, ε, διατροφική άλυσο. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι ο Ισπανικός νόμος βασίζεται σε μια κατάχρηση κυρίας και θέσης που στον κλάδο των τροφίμων και ιδιαίτερα των γαλακτοκομικών παρουσιάστηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα σκέφτομαι τη δική μου χώρα. Σήμερα πραγματικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα. Στην Ιταλία οργανώνονται πάρα πολλές διαδηλώσεις γιατί υπάρχει μια πολυεθνική η οποία έχει στα χέρια στην αγορά του νοπού γάλακτος. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πολυεθνική. Και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Πολύ δύσκολα οι φορείς στον τομέα αυτό θα μπορέσουν να αντλήσουν δυνάμεις για να μπορέσουν να, να κάνουν κάτι όχι μόνο για την αθέμητη πρακτική που θα τους επιτρέψει να αλλάξουν μονομερώς ε, τις, ε, ε, τα πράγματα στην αγορά. Το ερώτημα όμω που θέτω είναι η αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν εξουσία στην επιβολή συμβάσεων που κατά κάποιο τρόπο οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν ή να προσυποργάψουν και αυτό καθιστά δύσκολη τη θέση των κυβερνήσεων γιατί είναι δύσκολο το να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. Ε, συνεπώς το ερώτημα είναι η αποτελεσματικότητα και σε ό,τι αφορά την, ε, τις μεγάλες συμβάσεις που υπογράφονται με τις πολυεθνικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χαϊτέμα. Yes, thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολη γι' αυτό. Ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε. Πολύ ενημερωτική η παρουσίαση. Μια ερώτηση έμμεσα συναρτημένη με το θέμα σας. Θα τη θέσω λίγο ομά. Ξέρουμε ότι η μικροβιακή αντοχή είναι μεγάλο πρόβλημα. Εν μέρη προέρχεται από τις ζωοτροφές και τα φάρμακα που περιέχουν. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες, όπως ξέρουμε, που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, οι βουλευτές από την Ισπανία θέλουν να αποδυναμωθεί η νομοθεσία για τις ζωοτροφές με φάρμακα. Εσείς ως Υπουργός είστε υπέρ αυτής της άποψής τους ή ποια είναι η δική σας άποψη. Ε, πώς πιστεύετε ότι επηρεάζουν οι προσπάθειες των βουλευτών σας και πιστεύετε ότι πρέπει να χορηγείται αντιβίωση προληπτικά στα ζώα ως μια πρακτική, ε, ε, αφού είναι μια πρακτική που παραβιάζει και θέματα υγείας και κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Θα ήθελα η απάντηση ή δυνατόν να δοθεί και προφορικά και γραπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Σένορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ήμουν μία από τις συντονίστριες που ήταν κατά της παρουσίας σας εδώ σήμερα και της πρόσκλησης. Γιατί φανταζόμουν ότι θα παραλείπατε μερικά βασικά σημεία. Και όντως, δώσετε ως παράδειγμα το γαλακτοκομικό τομέα. Νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις που έγιναν το καλοκαίρι και η άρνηση δύο από τις τρεις οργανώσεις να υπογράψουν την τελική συμφωνία είναι μια περίτρανη αμφισβήτηση των υποτιθέμενων επιτυχιών που μας παρουσιάσατε από την εφαρμογή της σχετικής ισπανικής νομοθεσίας. Και βέβαια το δημόσιο σύστημα ρύθμισης ε, που μας παρουσιάσατε της επιστηστικής αλυσίδας παραλείπει ένα, ένα σημαντικό σημείο. Το θέμα της ε, τιμής ε, που θα πρέπει να ανταμείβει τον παραγωγό. Και αυτό το ξεχνάτε, γιατί όταν ρυθμίζετε, προβλέπετε σε νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν ε, ρυθμίζετε ούτε την παραγωγή, ούτε τις αγορές, ούτε το πώς επηρεάζουν τις αγορές οι κανόνες περί ανταγωνισμού. Απλώς εμποδίζεται να γίνει μια πραγματική διαπραγμάτευση της τιμής που ε, εισπράττουν οι παραγωγοί. Έτσι αυτές οι υποχρεωτικές συμβάσεις είναι ουσιαστικά ε, ένα νέο βαρύδιο, ένα καινούριο έρμα για, τη, για τους παραγωγούς, για τους κτηνοτρόφους, ε, που ξέρουν βέβαια πότε θα πληρωθούν, αλλά ξέρουν ότι η τιμή που θα λάβουν δεν είναι αυτή που τους, επιτρέπουν, ε, δεν είναι αυτή που τους επιτρέπει να ζήσουν από την παραγωγή τους. Ε, αμφισβητώ λοιπόν τις επιτυχίες σας και αμφιβάλλω για την ορθότητα αυτού του νόμου. Επίσης υπάρχουν διακλαδικές οργανώσεις στην Ισπανία. Εκεί εκπροσωπούνται όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας εφοδιασμού. Υπήρχαν και υπάρχουν γεωργικές ε, οργανώσεις ε, και γεωργικοί συνεταιρισμοί που εκπροσωπούν τους παραγωγούς ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους στην Ισπανία. Δεν χρειάζεται να εφεύρετε τίποτα, απλώς να ρυθμίσετε σωστά την κατάσταση για να έχουμε πραγματικές διαπραγματεύσεις ελάχιστης τιμής που θα επιτρέπουν το βιοπορισμό των γεωργών μας, των αγροτών μας και να επιτρέψουν την επιβίωση της γεωρικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Eh, Θα δώσω το λόγο στον καταναλώνο συνάδελφο τον κύριο Γιώργη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν ε, να συμπληρώσω και να, να πω στον εκπρόσωπο των φιλελευθέρων ότι δεν είναι όλοι οι Ισπανοί που συμφωνούν με αυτά που ακούσαμε. Έχετε δίκιο κύριε Υπουργέ ότι το γεγονός ότι επιτέλους έχουμε ένα νομοθέτημα βελτιώνει την προηγούμενη κατάσταση. Αλλά όπως είπε και η συνάδελφος ε, Σένερα, αν υπάρχει σαφής ε, μνήα του του δίκαιου τιμήματος που θα πρέπει να λαμβάνουν οι παραγωγοί αν δεν υπάρχει τέτοια ρητήμνια, ε, παραμένει χολή και ελλειπής αυτή η νομοθεσία. Μίλησατε για τον κώδικα καλών πρακτικών ε, της ε, αυτορύθμισης, αλλά δυστυχώς είναι προαιρετικός αυτός ο κώδικας. Όπως είπατε, μόνο οι εθελουσίες μπορούν να προσχωρούν σε αυτόν. Επίσης, ό,τι αφορά το, τα απορροκυπευτικά, η Ισπανία είναι χώρα εξαγωγή απορροκυπευτικών προϊόντων. Οπότε τα κρατικά μέτρα για τη βελτίωση της επιστημιστική αλυσίδας δεν ε, έχουν καμία ιδιαίτερη αξία για μια χώρα που εξάγει προ τι υπόλοιπε ευρωπαϊκές. Έχουμε μια οδηγία που προστατεύει τους ε, καταναλωτές από τις καταχρήσεις στην επισητιστική αλυσίδα. Αυτό όμως που μας προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των παραγωγών είναι και πάλι ένας απλός κώδικας βέλτιστων των πρακτικών και πάλι προαιρετικός, εκούσιος κώδικας. Το μεγαλύτερο τμήμα της απορροκυπευτικής παραγωγής που δεν μπορέσαμε να εξαγάγουμε προς τη Ρωσία λόγω του ρωσικού αποκλεισμού ε, με τους παραγωγούς να πληρώνουν τα σπασμένα ε, δεν κατευθυνόταν προς την ε, ευρωπαϊκή αγορά, αλλά προς την ισπανική αγορά. Οπότε χρειαζόμαστε κοινοτική νομοθεσία που θα προστατεύει ρητά όλους τους ε, ευρωπαίους παραγωγούς. Οι δεμοί τέτοιες ε, προαιρετικές απλώς ρυθμίσεις έχουν ελάχιστη αξία. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Ο κύριος Φεγόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εδώ μιλάμε για ένα νιωστή φορά, για ένα θέμα που αφορά τις ανισότητες που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μείωση των γεωργικών τιμών δεν είχε ανάμεση επίπτωση στους καταναλωτές θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ακούμε την άποψη κάθε χώρα μέλους για να γνωρίζουμε τα μέτρα που λαμβάνονται σε ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση. Αυτό όμως δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η επαρχή του προβλήματος βρίσκεται καταρχάς στην εφαρμογή μιας συμφωνίας η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τη μία ε, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη είναι σημαντικά στοιχεία αλλά έχει σχέση και με, το, με τις ίδιες τις τιμές. Χρειάζονται βεβαίως αποτελεσματικά μέσα για να ελεγχθεί η κυρίαρχη ε, θέση στον τομέα της διανομής. Θα ήθελα απλά και μόνο να σας πω ότι το μύθο θα πρέπει να μας απασχολήσουν είναι η συγκέντρωση των ε, συμφεροντούχων στον τομέα των ε, διατροφικών αγαθών. Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι πέρα από αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να ζητήσουμε τουλάχιστον μία επανεξέταση του δικαίου του ανταγωνισμού σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μαγκίνες, που όπως είπαμε είναι και συντάκτηρα της γραμμοδότησης ε, για τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Οι υπουργοί έρχονται συνήθως όταν προεδρεύουν στα συμβούλια. Γι' αυτό χαιρόμαστε που ήρθατε να μιλήσουμε για την εμπειρία σας και καλό είναι να γίνεται αυτό και με άλλους υπουργούς. Τρεις παρατηρήσεις είναι σαφείς. Ε, στην Ισπανία είδατε ότι χρειαζόταν ανάληψη δράσης και αναλάβατε πολιτική δράση. Γι' αυτό σας συγχαίρω. Δεύτερον, συνδυάσατε την νομοθεσία με την αυτορύθμιση, γιατί προς το παρόν σε επίπεδο ένωσης έχουμε ένα προαιρετικό εθελοντικό κώδικα την ε, πρωτοβουλία για την αλυσίδα τροφίμων. Έχουμε ένα κομμάτι όμως ε, ε, νομοθετικών προτάσεων που έχουμε σε επίπεδο ένωσης. Είναι σημαντικό να μπορούν να συνδυαστούν οι δύο προσεγγίσεις ε, επίσης ε, στην αρχή μιλήσατε για την ε, βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Εκεί εστιάζουμε. Αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι αυτή πρέπει να λειτουργεί. Και ο νόμος, η νομοθεσία περί ανταγωνισμού θα πρέπει και εκείνη να συνδράμει ε, ούτως ώστε να μην είναι χαλήνοτος ο ανταγωνισμός. Όπως και ο κύριος Ντες θα ήθελα πάρα πολύ ένα αντίγραφο της ομιλίας σας. Ε, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ήθελαν και γραπτά την ομιλία σας. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα ανησυχία σε σχέση με το νομοθεσία ανταγωνισμού. Ε, προήλθαν αντιστάσεις και από πού. Ε, και ποια είναι η φωνή των καταναλωτών, γιατί κάποιοι θα έλεγαν ότι θα πρέπει να λάβουν περισσότερο υπόψη τους καταναλωτές. Εγώ θεωρώ ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών δεν αποκλίνουν πολύ, ούτε είναι ασυμβίβαστο να ε, φροντίζουμε τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Ε, το λέω αυτό και στην έκθεσή μου, αλλά νομίζω ότι η παρουσίασή σας έδωσε άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και εδώ. Ευχαριστούμε. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι εγγράφονται στο κατάλογο των ομιλητών. Οπότε θα πρέπει να συντομεύουμε το χρόνο αγόρευσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, ε, επισκέπτες, ε, την ομάδα επισκεπτών του κυρίου Ντόρφμαν και να δώσω το λόγο στην κυρία Εράνς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την Ισπανίδα Υπουργό που ήρθε στην ε, συνεδρίαση και να συγχαρώ την Ισπανική κυβέρνηση για αυτή την πρωτοπόρο πρωτοβουλία που ανέλαβε και που απέφερε καρπούς. Φυσικά είναι βελτιώσιμη η πρόταση, αλλά ως πρώτο βήμα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και θετική πρωτοβουλία. Κύριε Υπουργέ, οι δυνατότητες βελτίωσης του νόμου ε, δεν θα διευρυνθούν αν γενικευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τέτοια πρωτοβουλία, ώστε να εξασφαλίσουμε ισορροπία μεταξύ όλων των κρίκων της επιστηστικής αλυσίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εθνικό. Γιατί έχουμε ενία αγορά. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε ισορροπία να υπάρχει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρίκων της αλυσίδας. Σε ό,τι αφορά τον γαλακτοκομικό τομέα, το γάλα θεωρώ ότι το, και το ευρωπαϊκό πακέτο για το γάλα είναι βελτιώσιμο. Το ίδιο και η επιρροή των οργανώσεων παραγωγών και οι ικανότητες που θα πρέπει να έχουν και οι δυνατότητες να επεμβαίνουν με πιο ισχυρό και αποφασιστικό τρόπο στην επιστηστική αλυσίδα. Δεν πιστεύετε ότι και το ευρωπαϊκό πακέτο για το γάλα θα πρέπει να ακολουθεί αυτή την άκουσα και να βελτιωθεί ριζικά. Επίσης, αυτός ο οργανισμός ε, ελέγχου και πληροφοριών, ΆΙΚΑ, στην Ισπανία, δεν είναι καλό παράδειγμα και για τις υπόλοιπες χώρες μέλη, ώστε όλες οι χώρες να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα παρατήρησης ε, και διερεύνησης της κατάστασης. Το ισπανικό παράδειγμα επίσης για την επιβολή σημαντικών οικονομικών κυρώσεων ε, δεν θα μπορούσαν να γίνει παράδειγμα προς και για τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Αν και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου μια και ε, είμαστε τρεις εβδομάδες ε, πριν τις εκλογές που θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου δεν είναι και ε, πρέπουσα η σημερινή παρουσία της Ισπανίδας Υπουργού, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν σε προεκλογική περίοδο, οπότε είναι αδόκιμη μια τέτοια εμφάνιση λίγο πριν τις εκλογές. Αυτά προκαταρκτικά και ως προς την ουσία. Είπατε ότι όταν αναλάβετε την εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια επικρατούσε χάος και χάρη σε εσά βελτιώθηκε η κατάσταση. Όχι, ούτε χάος υπήρχε πριν, ούτε εσείς ε, επιλύσατε διαμαγείας ε, τα προβλήματα των γεωργών και των κτηνοτρόφων της Ισπανίας. Ο νόμος αυτός μπορεί να είναι καλοπροαίρετος, να είναι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του νόμου είναι το συγκεκριμένο σύστημα κυρώσεων που θεσπίζει και η ίδρυση του Οργανισμού ε, για τον Έλεγχο και την Ενημέρωση του ΆΙΚΑ. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, η Κυρός και ο Άικα. Τώρα, ποιο είναι ο αδύναμο κρίκο τη αλυσίδα. Η παραγωγή, η και την οτρόφη. Οπότε θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα της, ε, των αγοροπολισιών χωρίς συμβάσεις και χωρίς καθορισμό τιμών. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί δεν ξέρουν οι παραγωγοί τι τιμές, ε, τι τιμή θα πληρωθούν για τα προϊόντα τους. Επίση, δύο σημαντικές βιομηχανίες, δύο σημαντικές επιχειρήσεις γαλακτοκομικές στην Ευρώπη ανανέωσαν τις συμβάσει τους ε, ε, με, με ισπανούς παραγωγούς, αλλά με πολύ μειωμένε τιμέ σχέση με το παρελθόν. Αυτή είναι η βελτίωση που ευαγγελιστήκατε. Επίση, ε, σε ό,τι αφορά τα έκτακτα μέτρα και την αύξηση της ποσόστοσης ελαιολάδου για την Τινησία, τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ε, και να πω στον ε, εκπρόσωπο των φιλελευθέρων ότι η άγνοια αποτελεί τη μεγαλύτερη θρασίτητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την επισκόπηση της κατάστασης. Χαίρομαι που δεν περιμένατε σπρόξιμο, αλλά να λάβατε την πρωτοβουλία και έχετε ήδη καλά αποτελέσματα. Ερώτηση. Δεν πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να είχαμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αντί για 28 εθνικά συστήματα που μπορεί να οδηγούν σε παραβιάσεις, ε, προσφυγές στη δικαιοσύνη, ε, συγκρούσεις. Νομίζω ότι ο γαλακτοκομικός τομέα αντιμετωπίζει το με μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και οι Λιθουανοί γαλακτοπαραγωγοί και καταναλωτές χθε μου υπέβαλαν έτοιμα με 40.000 4.500 υπογραφέ. αυτοί οι γαλακτοπαραγωγοί και οι καταναλωτές θέλουν να υιοθετήσουμε ενιαίο σύστημα με νέα συστήματα πληρωμών. <clears throat> Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε για να προλάβουμε κρίσεις μελλοντικέ και να φροντίσουμε ώστε οι αγρότες μας να μην ε, επομιστούν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η γαλακτοπαραγωγή και οι αγρότες να έχουν ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Εσείς τι λέτε για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τέτοιου ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος κατά των αθέμητων πρακτικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόστιγκερ. Äh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ερώτηση, συντομότατα. Εμείς ασχολούμεθα πάρα πολύ και με την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος και νομίζω ότι θα είναι απολύτως απαραίτητο να περάσουμε από το εθελεντικό σε ένα υποχρεωτικό σύστημα μέτρων. Αλλιώς οι, η ισχυροί στην, αγορά, στην αλυσίδα εφοδιασμού ε, δεν θα υποχωρήσουν. Ποια είναι η εμπειρία σας μετά τον νόμο στην Ισπανία, δηλαδή ποια δυνατά σημεία <clears throat> υπάρχουν, τι θα θέλατε εσείς να προσωπικά να βελτιωθεί και τι μπορούμε να συναγάγουμε ως συμπέρασμα για να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ένωσης. Θα ήθελα δηλαδή την εμπειρία σας αυτή να την αξιοποιήσουμε σε επίπεδο ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση σε ό,τι αφορά το χοιρινό κρέας. Επισκέφθηκα την Ισπανία και συζήτησα με πολλούς και μαθα ότι ένα κιλό χοιρινό κοστίζει λίγο περισσότερο από ένα ευρώ. Πώς καταφέρνετε να κρατήσετε ζωή αυτόν τον τομέα αφού το κόστος παραγωγής για ένα κιλό κρέατος είναι περίπου το ίδιο με την τιμή πώλησης. Υπάρχουν μηχανισμοί που επιβάλλονται από την κυβέρνηση και βοηθούν τους ε, κτηνοτρόφους να επιβιώσουν γιατί πραγματικά δεν, καταφέ, δεν καταλαβαίνω πώς καταφέρνουν να, επιβιώσουν αφού η τιμή παραγωγής είναι η ίδια με την τιμή πώλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ήδη διατυπώθηκε η ερώτησή μου. Παρ' όλα αυτά την επαναλαμβάνω. Στην Ισπανία και τον δικό σας τρόπο προσέγγιση από την νομική άποψη θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομική προσέγγιση ή νομίζετε ότι θα δημιουργούσε προσκόμματα. Δηλαδή το να υπάρχει επιπλέον νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δυσκόλευε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλάβαμε με την παρέμβαση της κυρίας Υπουργού Παρίνη προσέγγιση της Ισπανίας. Πιστεύω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα καταφέρουμε ή δεν θέλουμε να μάθουμε από αυτή την εμπειρία. Χαίρομαι όμως που η χώρα σας πραγματικά έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Η προσέγγιση γίνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Υπάρχει ένας νόμος που συνδέεται με ελέγχου και με κυρώσει, δηλαδή έχει κατασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία, καλύτερες εμπορικές τιμές, καλύτερη ρύθμιση των διαφορών ε, και σήματα κινδύνου στο ίδιο το σύστημα. Σε αυτή την ε, αλυσίδα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπλοκή όχι μόνο των άμεσα ενδιαφερομένων αλλά και των καταναλωτών ο γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από το μονοπόλιο μεγάλων επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν στο δημόσιο σύστημα όπως προβλέπετε από τον νόμο σας να υπάρχει η συμμετοχή και των καταναλωτών. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτό το τομέα και ελπίζω ότι η εμπειρία της Ισπανίας θα βοηθήσει και τις άλλες χώρες. Είναι σαφές ότι ένας και μοναδικός νόμος δεν, θα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε χώρας. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν επιθυμητή μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. ευχαριστώ κύριε Oui, merci, le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την ε, παρουσίασή της. Είναι αλήθεια ότι ενώπιον ενός προβλήματος τουλάχιστον εσείς κάνατε κάτι και προσπαθήσατε να βρείτε απαντήσεις καταλαβαίνοντας ορισμένα στοιχεία και περιορισμούς. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι αυτά. Θα βλέπει να δούμε αν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση win-win. Εδώ το θέμα των τιμών που τίθεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος ορίζει τις τιμές, πώς ορίζονται οι τιμές. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κάθε χρόνο πολλά ζώα και τάβροι συγκεκριμένα ε, πεθαίνουν υποφέροντας φρικτά βάσανα στις αρένες της Ισπανίας και πολλά χωριά κάνουν γιορτές με βαρβαρικά έθιμα ε, όπως την Τούρα όπου ε, έφυποι σκοτώνουν τους σταύρους ε, με κοντάρια και έχουμε και το Κόρτε Βίγκο που θα γίνει σύντομα και εκεί ε, βάζουν φωτιά στους σταύρους και τους κυνηγούν. Πολλοί Ευρωπαίοι και οι περισσότεροι Ισπανοί πολίτες θέλουν αυτά να σταματήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να τερματίσει τις σταυρομαχίες και θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε την ε, παραγωγή, την εκτροφή αυτών των ταύρων. Ε, είναι τρομερές, είναι φρικαλές αυτές οι πρακτικές. Ε, πρέπει να λάβετε υπόψη και τις απόψεις των πολιτών που θέλουν να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστώ. Κύριε Σκούσμιουκ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Έχω δύο ερωτήσεις. Ο νόμος αυτός ισχύει στη Ισπανία εδώ και ένα χρόνο και. Οπότε μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια ήταν τα αποτελέσματά του και πώς επηρέασε τα γεωργικά εισοδήματα. Χάρη στην εφαρμογή του νόμου αυτού βελτιώθηκαν τα γεωργικά εισοδήματα. Επίσης, πώς επηρέασε η εφαρμογή των, του νόμου τις τιμές του καταναλωτή. Υπήρξε κάποια αύξηση των τιμών μετά την εφαρμογή και τη θέση ίσχυ του νόμου. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό ελέγχου και ενημέρωσης που είπατε ότι επιβλέπει την κατάσταση και μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Έχουν ήδη εφαρμοστεί κυρώσεις ε, και αν ναι, τι ύψους ήταν οι χρηματικές ε, ποινές που επιβλήθηκαν. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρτίνες. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που ήρθατε. Παρόλο που σίγουρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή, ε, δεδομένου ότι επίκυνται εκλογέ στην Ισπανία. Έχουμε τον νόμο λοιπόν ε, για την επιστημιστική αλυσίδα που είναι γεμάτος κενά και ατέλειες. Πώς μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι βελτιώνει την κατάσταση των γεωργών και κτηνοτρόφων αν έχει, αφού, από τη στιγμή που έχει μειωθεί το εισόδημά τους κατά 7,1%. Ζούμε επίσης ε, τις χειρότερες χρονιές για τους γαλακτοπαραγωγούς στην Ισπανία. Φαίνεται ότι ζούμε σε διαφορετικές χώρες κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι αρκούν οι κυρώσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Πιστεύετε ότι χρειάζεται απλώς κυρώσεις ή να αλλάξουμε ολόκληρο το μοντέλο ώστε να προστατεύσουμε τους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας για να δώσουμε πραγματικά αξία και να αναβαθμίσουμε το έργο τους. Ευχαριστώ κύριε Σάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί καθημερινά στις συναντήσεις μας. Σήμερα έχουμε μια συνάντηση με 200 κτηνοτρόφους Ολλανδούς. Έγιναν και συγκεντρώσεις στις Στη χώρα σας ανασκουμποθήκατε από ό,τι κατάλαβα. Ο Βέλγος Υπουργός και η Οργάνωση Γεωργών στο Βέλγιο υπέβαλαν πάρα πολύ καλά προγράμματα και ιδέες. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει μία λύση σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως και η διάσταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση η γεωργή της εκλογικής μου περιφέρειας. Έχασαν κονδύλια μολονότι είχαν συνεργαστεί μέσα, μαζί, μεταξύ τους στα πλαίσια συνεταιρισμών. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρέμβασή της, αλλά και για τη σημερινή της παρουσία. Θα ήθελα να εκφράσω έναν προβληματισμό καταρχάς, να τη συγχαρώ την Ισπανική κυβέρνηση για την πρωτοβουλία της Βεβαίω ε, δεν έχουμε ακόμα κάποια ανατροφοδότηση για να ορίζουμε το πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά. Παρόλα αυτά υπάρχει μια βέλτιστη πρακτική που θα πρέπει να συναγωνιστούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ελπίζω λοιπόν ότι σύντομα θα μπορέσει να υπάρχει ένας εναρμονισμένος, μια εναρμονισμένη νομοθεσία. Παρατηρώ ότι ο Υπουργό δύο φορές αναφέρθηκε στο θέμα της απάτης ε, στο διατροφικό τομέα. Ενδεχομένως αυτό είναι το θέμα των θεμάτων στην Ευρώπη. Και θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να μου πείτε πώς και σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, οι ευρωπαϊκές διαδικασίες για να υπάρξει ένας εντοπισμός των απατών σε ό,τι αφορά την ετικετοθεσία και την ονομασία προέλευσης ειδών διατροφής. Εξαντλήσαμε το κατάλογο των αγορητών. 23 ε, συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο και υπέβαλαν ερωτήσεις. Έχω κι εγώ μία ερώτηση. Έχετε παρουσιάσει το νόμο αυτό στο Συμβουλίο Υπουργών γιατί φαντάζομαι έχετε συζητήσει επανειλημμένω για το θέμα αυτό. Έχετε παρουσιάσει όπως το κάνατε σε εμά τον νόμο σας στους συναδέλφους σας, Υπουργούς Γεωργίας, στο Συμβούλιο. Ακούσατε, κυρία Υπουργέ, πληθώρα ερωτήσεων. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε διεξοδικά σε όλες. Ε, έχετε το λόγο και σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τους ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις τους και τις ερωτήσεις τους. Μερικές βέβαια ήταν πολύ μακριά από το θέμα του νόμου για την βελτίωση της λειτουργίας της επιστηστικής αλυσίδας που ήταν και το αντικείμενο της πρόσκλησης, ενώ μερικά σχόλια ήταν εκτός θέματος. Εν πάση περιπτώσει. Με ρωτήσετε πώς δέχθηκαν οι αλυσίδες διανομής της κυρώσης και τι έγινε με τα απορροκυπευτικά, αν τις δέχτηκαν εύκολα ή με βαριά καρδιά. Βέβαια, οι οι φορεί τη διανομή είχαν πολύ, ισχυρή διαπραγματευτική, πολύ μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ πριν την εφαρμογή του νόμου. Κάτι που ίσχυε και στις υπόλοιπες και ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα να καρπώνονται μεγάλο τμήμα της αξίας της διαπιστιστικής αλυσίδα βάρος ε, των παραγωγών. Όπως είπα στην αρχή, το νομοθέτημα αυτό είναι για όλους και υπερπάντων. Θέλουμε να ενισχύσουμε όλους τους κρίκους αλυσίδας από την πρώτη στιγμή εμπλέξαμε και τους διανομής στη διαδικασία με τους υπόλοιπους φορείς και καταλήξαμε σε ένα πολύ φιλόδοξο νομοθέτημα που εκπονήθηκε με τη συμφωνία και της ε, διανομής και του κλάδου της διανομής. Ε, κατάλαβαν ε, οι εταιρείε της διανομής ότι έπρεπε να αλλάξουν τις πρακτικές τους και γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση τους παρότρινε και η Ισπανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ε, ο νόμος αυτός έτυχε και της αποδοχής ε, του κλάδου της διανομής. Σε ό,τι αφορά το κώδικα βέλτιστων των πρακτικών, όντως είναι εθελοντικός, καθυστερήσαμε δύο χρόνια για την εισαγωγή του. Ναι, μεν είναι προαιρετικός, αλλά παρόλα αυτά πολλοί έχουν προσχωρήσει ήδη στον κώδικα αυτό. Χρειάστηκε κόπος και χρόνος, αλλά τελικά πολύ προσχώρησαν, γιατί φυσικά όντω μια προαιρετική ρυθμίση δεν έχει νόημα αν ε, οι ενδιαφερόμενοι δεν ε, την εφαρμόζουν. Επαναλαμβάνω όμω και ο κώδικας έτυχε τη σύμφωνη γνώμη των φορέων και της διανομής. Μιλήσατε για το, τα απορροκυπευτικά κυρίως και τι προθεσμίε. Υπάρχει ένα σχέδιο αυτεπάγγελτων ελέγχων εκ μέρου του Οργανισμού Ελέγχου και ενημέρωση. Είναι ένα, ένα σύστημα που βρίσκεται εν εξελίξη, δεν είναι καθόλου στατικό. Προσαρμόζεται στις περιπτώσεις. Και όταν ξεκίνησε πέρυσι αυτό το σύστημα ελέγχων, επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στον τομέα των περικυπευτικών, γιατί ακριβώς λόγω του ρωσικού αποκλεισμού χάθηκε ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς, ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Και σκεφτήκαμε ότι ίσως έτσι ο κλάδος βρεθεί σε πολύ πιο ευάλωτη θέση. Γι' αυτό και ενισχύσαμε ιδιαίτερα τους ελέγχους στον τομέα των απορροκυπευτικών σε όλους τους κρίκους της επιστηστικής αλυσίδας. Το ίδιο ισχύει και με το γάλα. Και ο γαλακτοκομικός τομέας ε, αντιμετωπίζει προβλήματα στην Ισπανία, κάτι που δεν εξαίρεσε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και η έλεγχη στο γαλακτοκομικό τομέα είναι πιο ενισχυμένη. Δίνουμε προτεραιότητα στο γαλακτοκομικό τομέα εξαιτία των αντίξεων συνθήκων που ισχύουν αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έλεγχοι του οργανισμού ΑΕΚΑ, του Οργανισμού Ελέγχου και Ενημέρωση, επαναλαμβάνω, έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα και αλλάζουν ανάλογα με τι ανάγκε ε, και ανάλογα με τι περιπτώσει και την ε, τροτότητα που παρουσιάζει ο Α ή Β Σίγουρα θα σας ε, στείλω την ε, ομιλία μου από τη στιγμή που τη ζητήσατε. Εκεί θα δείτε μεγαλύτερες, περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τα πέντε σημεία, τα πέντε επιμέρους σημεία του νόμου, αλλά αν δεν αρκεί η ομιλία που απλώς ακροθυγώς αναφέρεται στα σημεία αυτά, μπορώ να σας στείλω και πολύ μεγαλύτερες νομικές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του νόμου. Ο κύριος Δεκάστρο μίλησε για την αποτελεσματικότητα του νόμου σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ε, εταιρείες, ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα. Κάποια, ε, κάποιες πρακτικές που θεωρούνταν συνηθισμένες τώρα πια έχουν χαρακτηριστεί αθέμητες ε, και τιμωρούνται. Μάλιστα πριν την σύναψη σύμβασης θα πρέπει να συντρέχουν έχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να ε, είναι ανεξέλεγκτες οι συμβάσεις. Θα πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Και ο νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, άσχετα με το μέγεθός τους. Και ιδιαίτερα εφαρμόζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση και μερικές φορές και σε δεσπόσα θέση. Ακριβώς ε, Γι' αυτό λοιπόν οι κυρώσεις που επιβάλλουμε κυρίως ε, επιβάλλονται σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ροπή προς τις καταχρήσεις. Και ο νόμος ορίζει τις αθέμητες και καταχρηστικές πρακτικές. Γι' αυτές επιβάλλονται κυρώσεις και για τις συμβάσεις υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός προϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν ε, για τις ε, συμβάσεις. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις επιβάλλονται κυρώσεις. Κάποιος μίλησε για τη μικροβιακή αντοχή. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο ε, του νόμου για τη βελτίωση της λειτουργίας της επιστημιστικής αλυσίδας. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι η Ισπανία εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα για, την, ε, για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής, ε, κάτι που κάνουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες φαντάζομαι. Εμείς στηρούμε την ενωσιακή νομοθεσία και ας μην μπερδεύουμε τη μικροβιακή αντοχή των ζώων με τον τρόπο χορήγησης ε, των φαρμάκων στα ζώα. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση αυτή δεν είναι του θέματος σήμερα ε, εκπίπτει του πεδίου εφαρμογή του νόμου. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε τη χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά άλλη χορήγηση των ε, φαρμάκων ή των αντιβιωτικών. Επαναλαμβάνω, η Ισπανία εφαρμόζει πιστά όλα τα μέτρα για, την, για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής, όπως προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία. Η κυρία Σένερα μίλησε για το γάλα και για την ευρωπαϊκή κρίση που διανύει ο κλάδος. Η κρίση του γάλακτος είναι πανευρωπαϊκή, δεν είναι μόνο ισπανική. Και μάλιστα η συνέπειε τη Ισπανία ήταν διαφορετικέ. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται εξαρτάται η κρίση και η οξύτητά της από το βαθμό ε, οργάνωσης των γαλακτοπαραγωγών. Εμείς προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες του γαλακτοκομικού τομέα και ε, ο νόμος αυτός ωφέλησε κυρίως ε, το γαλακτοκομικό τομέα πολύ περισσότερο στην Ισπανία από τις άλλες χώρες που δεν ίσχυε αντίστοιχη νομοθεσία το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση μας ήταν να προστατεύσει την κοινή γεωργική πολιτική, όχι μόνο με τον προπολογισμό που είναι 47 δις, που είναι πολύ μεγαλύτερο για την επόμενη περίοδο από ό,τι για την προηγούμενη 2007-2013, αλλά εμεί ταχθήκαμε υπέρ μια μεταρρύθμιση κοινή γεωργική πολιτική με τρόπο που να ευνοεί το γαλακτοκομικό τομέα. Ήμασταν κατά της, ε, του φόρου στο γαλακτοκομικό τομέα. Ε, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν επιζήμιο, παρόλο που δεν υπήρχε συμφωνία στο Συμβούλιο και μάλιστα 15 ε, εκατομμύρια ευρώ αφιερώσαμε φέτος από το αποθεματικό μας για το καλακτοκομικό τομέα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και μάλιστα διατηρήσαμε κάποιες ενισχύσεις που είναι 500 ευρώ το εκτάριο για το καλακτοκομικό τομέα, ενώ 229 είναι για τους υπόλοιπους παραγωγούς. Επίσης με τις συνδεδεμένες πληρωμές προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη ε, τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Γι' αυτό και αυξήσαμε κατά 50 κατά 56% τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στον γαλακτοκομικό τομέα. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες από το, τέλος από το πέρας των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Εγώ ανέκαθεν ε, ήμουν υπέρμαχο του καλακτοκομικού τομέα και είπα ότι άσχετα με τη συγκυριακή κατάσταση των τιμών, σε καμία περίπτωση θα πρέπει να κλείσουν εκμεταλλεύσει. Και δήλωσα ότι θα εφαρμόσουμε όλα τα νόμιμα μέτρα και σε εθνικό επίπεδο και θα υποστηρίξουμε αντίστοιχα μέτρα και σε κοινοτικό επίπεδο. Και ζητήσαμε τη συνεργασία του συνόλου των κρίκων της ε, επιστηστικής αλυσίδας ε, για την προστασία των κτηνοτρόφων. Επίσης η Ισπανία ε, διαπραγματεύτηκε 25 ε, συν 5 ε, εκατομμύρια για τον τομέα αυτό και είχαμε και πολλά εθνικά μέτρα. Στηρίξαμε και τις ενώσεις παραγωγών. Επίσης προβλέψαμε και εθνικά μέτρα για την πρόθεση της κατανάλωσης του γάλακτος πέραν των κοινοτικών και Επαναλαμβάνω, έχουμε ειδικά μέτρα στο νόμο αυτό για το γαλακτοκομικό τομέα. Ε, διευκόλυνση των πιστώσεων ε, και της πρόσβασης ε, στα δάνεια των κτηνοτρόφων. Δώσαμε ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη διαπραγματευτική ισχύ στις διακλαδικές οργανώσεις των κτηνοτρόφων. Προωθήσαμε την κατανάλωση του γάλακτος στα σχολεία. Έχουμε πολλά μέτρα ανάπτυξης πέθρου εκπονούμε ένα στρατηγικό σχέδιο για το γαλακτοκομικό τομέα. Πραγματικά, ε, ακριβώς επειδή είμαστε σε πολύ πίσω σε σχέση με την οργάνωση των παραγωγών, προωθούμε τα μέτρα ε, οργάνωσης των κτηνοτρόφων και θεσπίσαμε και 7 επιπλέον μέτρα με 31 εκατομμύρια ευρώ με άμεση ενίσχυση 30 ευρώ ανά αγελάδα. Έτσι οι περισσότερες ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις ε, θα υποφεληθούν και κυρίως στη Γαλλικία. Επίσης έχουμε για ένα χρόνο πάγωμα των πιστώσεων από το Υπουργείο. Έχουμε βελτιώσει λοιπόν και με σχετικό διάταγμα την εύρυθμη λειτουργία της επιστηστικής αλυσίδας ιδιαίτερα για το γάλα. Θέλουμε να έχει βιωσιμότητα ο γαλακτοκομικός τομέας. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν τάσσονται υπέρ της προστασίας του γαλακτοκομικού τομέα. Φυσικά στα πλαίσια της στρατηγικής μας ε, πολιτικής και για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα πολλά μέτρα που έχουμε προβλέψει για το γαλακτοκομικό τομέα και από οικονομική άποψη φέτος ε, έχουμε κινητοποιήσει πάνω από 800 ε, επιπλέον εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 200 που είχαν αρχικά αφιερωθεί στον κλάδο. Προσπαθούμε έτσι να βελτιώσουμε την κατάσταση με αυτή τη σημαντική ένεση ρευστότητα των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Από την αρχή ταχθήκαμε υπέρ του γαλακτοκομικού ε, πακέτου, ζητήσαμε υποχρεωτικές συμβάσει και ενισχύσαμε τις οργανώσεις παραγωγών. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε πείρα και δώσαμε μεγαλύτερη ισχύ στι οργανώσει παραγωγών ε, με μεγαλύτερε απαιτήσει για την εφαρμογή των συμβάσεων. Μην ξεχνάτε ότι εκτός ότι ρυθμίσαμε την υποχρέωση σύναψη σύμβασης, έχουμε ένα σύστημα που προβλέπει και κυρώσεις. Αυτό προβλέπει ο νόμος μας. Βέβαια, οι υπόλοιπε χώρε δεν εφαρμόζουν υποχρεωτικά συμβάσει. Από ό,τι ξέρω, καμία άλλη χώρα πλην τη Ισπανία ε, δεν έχει σύστημα ε, επιβολή κυρώσεων προκειμένου να ελέγχει την πραγματική εφαρμογή τη υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Αν όλα αυτά δεν προστατεύουν του γαλακτοπαραγού στην Ισπανία, τι, τι άλλο κάνει. Τι άλλο θα μπορούσε να το κάνει. Επαναλαμβάνω, δίνουμε ενάψματα και για την ε, οργάνωση, την καλύτερη οργάνωση των ε, παραγωγών. Με όριο μάλιστα 33% για την εκπροσώπηση. Κάτι που προβλέπεται και στην κοινωτική νομοθεσία. Από αυτή την άποψη, ο πιο προστατευμένος τομέας στην Ισπανία είναι ο γαλακτοκομικός τομέας. Οι στην Ισπανία. Ο κύριο Σεμπαστιά μίλησε για μια ελάχιστη τιμή, για μια κατώτατη τιμή. Πιστεύω ότι θα πρέπει κυρίω να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών. Τώρα να μιλούμε για ελάχιστη τιμή, αυτό δεν μα το επιτρέπει η ιδρυτική συνθήκη τη Ένωση και αντιβαίνει στου κανόνε του θεμετού ανταγωνισμού αλλά και στην ισπανική νομοθεσία. Δεν μπορούμε να μιλούμε για κατώτατη τιμή, για εξασφάλιση κατώτατης τιμής. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στο κοινοτικό κεκτημένο. Μιλήσαμε και για τον κώδικα καλών εμπορικών πρακτικών. Είπατε ότι δεν αρκεί γιατί έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Μπορεί να μην ε, με καταλάβατε γιατί ο νόμος απαρτίζεται από πέντε σημεία. Ένα ήταν το υποχρεωτικό, η διοικητική ρυθμίση και ένα ήταν το προαιρετικό, η αυτορυθμίση. Υπάρχει και ένα τμήμα που είναι υποχρεωτικό. Μην εμένετε μόνο στο προαιρετικό. Το υποχρεωτικό τμήμα περιλαμβάνει και κυρώσεις και μάλιστα συστήσαμε ειδικό οργανισμό που εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και έχει και την ικανότητα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο κώδικας των πρακτικών είναι μόνο ένα τμήμα του νόμου που ξεπερνάει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του δημόσιου σκέλους ε, του υποχρεωτικού. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι ή εθνικές ρυθμίσεις ε, μόνο της Ισπανίας. Ο κύριος Φεράν μίλησε για τη συγκέντρωση των εμπορικών τελεστών, ε, κυρίως ε, στον κλάδο της διανομής. Αυτό είναι κάτι προφανές που εμφανίζεται και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε την συγκέντρωση και την οργάνωση των παραγωγών. Στην Ισπανία υστερούμε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες ό,τι αφορά την οργάνωση της οργανώση των παραγωγών. Δεν έχουν αυτή την οτροπία της οργάνωσης, αυτή την προωθούμε. Επίσης με την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, όχι μόνο στο γαλακτοκομικό τομέα και μέσω της προώθησης των διακλαδικών οργανώσεων, ε, δίνουμε έμφαση στην ανάγκη οργάνωσης και επίσης ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε του συνεταιρισμού ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθο και βαρύτητα και να διαπραγματεύονται ίσω προ ίσω με τον κλάδο τη διανομή. Μάλιστα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Πέθρου προβλέπουμε 226 επιπλέον εκατομμύρια για να ενισχύσουμε τις, τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών και άρα να αυξήσουμε τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Η κυρία Μαγκίνες μίλησε για την ε, ανάγκη τροποποίησης ε, των διατάξεων ε, περί ανταγωνισμού. Ο γαλακτοκομικός τομέας ε, είναι εξαίρεση με αυτό το 33% που προβλέπει. Εμείς εξαντλήσαμε τις δυνατότητες της κοινοτικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Μάλιστα το νόμο το διαπραγματευτήκαμε με το Υπουργείο Οικονομικών και με τη βοήθεια της Ισπανικής Αρχής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, νομίζω ότι η λιγότερη προστασία για τους καταναλωτές θα ήταν ένας ανεξέλεγκτος ε, κλάδος των παραγωγών ε, ή να αφήσουμε τους παραγωγούς στο έλεος της διανομής. Υπάρχει ένα πλέγμα διατάξεων ε, οικονομικών, περιβαλλοντικών και εθνικών και εθνικών και κοινοτικών Οπότε το, χειρότερο, το μεγαλύτερο κακό για τους καταναλωτές θα ήταν μια υποβάθμιση των κανόνων και των προδιαγραφών μας. Αν αφήσουμε εκτεθειμένους τους παραγωγούς, ουσιαστικά αφήνουμε και τους καταναλωτές απροστάτευτους. Θέλουμε μια ισορροπημένη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμό με ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις. Αυτό θα ωφελήσει όλους τους κρίκους αλυσίδα. Και μπορεί η ισορροπία των κρίκων της αλυσίδα να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει τους παραγωγούς. Και θα βοηθήσει, θα ενισχύσει την διαπραγματευτική του ισχύ με τον κλάδο διανομής. Φυσικά επιδέχεται βελτιώσει ο νόμος και φυσικά θα είμαστε υπέρ της Αντίστοιχη εφαρμογή μέτρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπατε είναι σχετικά νέος αυτός ο κανόνας, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ελεγχθεί η εφαρμογή του και χάρη στο παρατηρητήριο θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για να αποκτήσουμε καλύτερη επισκόπηση της επιστηστικής αλυσίδας και στην πορεία θα δούμε τι βελτιώσεις χρειάζονται. Ο ίδιος ο νόμος προβλέπει τρόπους βελτίωσής του. Τώρα, αν με την ε, εφαρμογή κάποιων ευρωπαϊκών μέτρων θα βελτιωθεί ε, ο νόμος, σίγουρα είμαι υπέρ αντίστοιχης θέσπισης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες που κάνει για την πάταξη των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και μάλιστα η πρόσκληση που μου απευθύνεται δείχνει την βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλλει στην ανέβρεση κοινών λύσεων για αυτά τα προβλήματα που μαστίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και το πιο ενδεδειγμένο επίπεδο για την ανέβρεση λύσεων είναι και το ευρωπαϊκό. Εγώ απλώς σας παρουσίασα την ισπανική εμπειρία. Είναι το δικό μας λιθαράκι στη συζήτηση. Πάντως όσο περισσότερο προχωρούμε προς ένα κοινοτικό σύστημα, τόσο περισσότερο θα προστατεύσουμε τους εμπορικούς μας τελεστές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε μία ενιαία αγορά. Και εκεί οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των φορέων και μεταξύ των κρατών μελών είναι συνεχής. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε κοινοτική λύση. Αυτό το είπα και στην αρχή. Σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, το είπα προηγουμένω, επ' ευκαιρία του γαλακτοκομικού τομέα. Στην Ισπανία η κτηνοτρόφη είναι η πιο προστατευμένη παραγωγή. Γιατί ο νόμος ακριβώς ε, εφαρμόστηκε προκειμένου να προσθέσει και ένα καθεστώς κυρώσεων σε περίπτωση που παρατηρούνται αθετήσεις ή μη συμμόρφωση με την υποχρεωτικότητα των συμβάσεων και η ύπαρξη του Οργανισμού Ελέγχου και Ενημέρωσης αποτελεί κλειδί στην εφαρμογή του νόμου. Γιατί ένας νόμος που απλώς απαγορεύει αλλά δεν τιμωρεί είναι απλώς μια δήλωση αγαθών προθέσεων. Είναι μια διακήρυξη προθέσεων, ένα ευχολόγιο ή ένας κατάλογος συστάσεων. Αν δεν έχουμε αντίστοιχο σύστημα επιβολής κυρώσεων, μένει αδύναμος ε, ο νόμος. Αυτό λοιπόν τον ε, χαρακτήρα της επιβολής των κυρώσεων έχει ο σχετικός οργανισμός ελέγχου και ενημέρωσης. Απαραίτητο συμπλήρωμα του νόμου και έχει έγκυο της ισχύω του. Και μάλιστα έχουν ένα προοδευτικό χαρακτήρα οι κυρώσεις, ε, στο μέτρο που οι παραβιάσεις έχουν ε, εξακολουθητικό χαρακτήρα, οι κυρώσεις γίνονται και πιο αυστηρές. Η κυρία Γιλέρα μίλησε για τις αγοραπολισίες σε τιμή κάτω του κόστους και τις ζημίες που επιφέρει κάτι τέτοιο για τους παραγωγούς. Ο νόμος 7 του 1996 ρυθμίζει το θέμα των αγοραπολισιών σε τιμές κάτω του κόστους. Δεν είναι αντικείμενο του τελευταίου νόμου που σας παρουσίασα. Οι πωλήσει με ζημίες κάτω του κόστους, επαναλαμβάνω, αποτελούν αντικείμενο άλλου νόμου. Πολλές καταγγελίες γίνονται στον οργανισμό ΆΙΚΑ και εμείς παραπέμπουμε το θέμα στις αυτόνομες διοικήσεις. Αυτές έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση που γίνονται πωλήσει κάτω του κόστους αλλά αυτό αποτελεί το αντικείμενο του νόμου για το λιανεμπόριο, του νόμου 7 του 1996. Σε περίπτωση που υπάρχουν σχετικές καταγγελίες, παραπέμπουμε το ζήτημα αυτό στις, στην τοπική διοίκηση. Ε, μιλήσατε για την ποσόστοση, τη διεύρυνση της ποσόστοσης ελαιολάδου για την Τινησία. Εμείς ταχθήκαμε κατά του μέτρου αυτού στο Συμβούλιο Υπουργών και εμείς ε, ζητήσαμε με δύο προτάσεις ε, ε, την αποθεματοποίηση ελαιολάδου, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, γιατί είχαμε πολλά πλεονάσματα και πέρυσι είχαμε 1.100.000 τόνους επιπλέον. Οπότε δώσαμε μάχη όχι μόνο για ε, τον γαλακτοκομικό τομέα, αλλά και για τον τομέα ελαιολάδου. Και ταχθήκαμε και κατά του σχετικού φόρου, του δασμού μάλλον, γιατί θα οδηγούσε σε τεράστιες ζημιές για τους παραγωγούς. Οπότε διαπραγματευτήκαμε τα 47 επιπλέον δισεκατομμύρια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη γεωργία. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία με τον κλάδο για να βρούμε διέξοδο για την εμπορία των προϊόντων. Γιατί το 2012 που είχαμε ιδιωτική αποθεματοποίηση καταφέραμε φέτος μέσα σε λίγα χρόνια δηλαδή, μέσα σε τρία χρόνια να διοχετεύσουμε σχεδόν ολόκληρη την παραγωγή. Κύριε Κιώστιγκερ μίλησε για ένα ενοποιημένο καθεστώς για τον γαλακτοκομικό τομέα Όντως, όταν έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ 28 χωρών μελών, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η Ισπανία αποφάσισε να εφαρμόσει από την αρχή το γαλακτοκομικό πακέτο και μάλιστα να το τελειοποιήσει. Και οι οργανώσεις παραγωγών έχουν πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σε αλυσίδες διανομής από τους μεμονωμένους παραγωγούς. Γι' αυτό και ενισχύσαμε την οργάνωση των παραγωγών. Αλλά και η συζήτηση για το γαλακτοκομικό πακέτο θα είναι πολύ σημαντική. Και καλό θα, γίνει, καλό θα είναι να, γίνεται, να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο για να προστατεύσουμε καλύτερα το γαλακτοκομικό τομέα από τις ανισορροπίες είτε στην κοινοτική είτε στην παγκόσμια αγορά. Είπατε ότι ο νόμος είναι ατελής και τι μπορεί να διδαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αδυναμίες του. Είναι πολύ νωρί για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα του νόμου. Εγώ θεωρώ ότι είναι καινοτόμο και πρωτοπόρο. Χρειαζόμαστε χρόνο όμω για να τον αποτιμήσουμε. Εγώ σα παρουσίασα τη μέχρι τώρα εμπειρία μα, αλλά καλό θα ήταν να περιμένουμε λίγο ακόμη για να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι. Μιλήσατε για την τιμή χείριο κρέατος, ένα ευρώ είπατε στην Ισπανία το χείριο κρέας κοστίζει 1,60 ευρώ. Δεν ξέρω που βρήκατε την πληροφορία αυτή για 1 ευρώ μόνο το κιλό για το χείριο κρέας. Ο, χείριος, ο τομέας χείριου κρέατος στην Ισπανία είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και μάλιστα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες ε, υγειονομικού ή οικονομικού χαρακτήρα, αλλά καταλήξαμε σε ένα επίπεδο ολοκλήρωσης ε, επαγγελματισμού και συγκέντρωσης ε, που μας ε, επέτρεψε να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάποιος άλλος ευρωβουλευτής μίλησε για την ανάγκη ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο. Και εγώ τάχτηκα υπέρ αυτής της κοινοτικής ρύθμισης και σίγουρα εδώ θα συμβάλλει ιδιαίτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις δικές του εργασίες. Μια και έχουμε ενιαία αγορά και εμπορικές συναλλαγές προς όλες τις κατευθύνσεις, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκές, δεν μπορούν να περιορίζονται σε εθνικά μέτρα. Για τους καταναλωτές, μίλησα προηγουμένως για το ρόλο των καταναλωτών. Οι οργανώσεις των καταναλωτών συμμετείχαν από την αρχή στο σχεδιασμό, εκπόνηση και θέσπιση του νόμου και συμμετέχουν και στο παρατηρητήριο για την επιστηστική αλυσίδα. Συμμετείχαν άλλωστε και στις εργασίες του κώδικα θεμητών εμπορικών πρακτικών. Με την εφαρμογή του νόμου δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Η αύξηση των τιμών οφείλεται στη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Εμείς απλώς θέλησαμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων κρίκων της. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των τιμών, πέραν τους μηχανισμούς παρέμβασης που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, και οι κανόνες του ανταγωνισμού, θα πρέπει να τους στηρίσουμε. Αυτό προβλέπει και ο νόμος. Και ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα και ως προς την εξισορρόπηση της διαπραγματευτικής ισχύω. Γιατί στις εμπορικές εναλλαγές μια ισότιμη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων καταλήγει και πιο σε ισορροπημένες τιμές, γιατί δεν έχουμε πια δεσπόζουσες θέσεις στην αλυσίδα επισητισμού. Τώρα για τις ταυρομαχίες και τους Σταύρους τις ενισχύσεις ε, της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, τις λαμβάνουν ε, μόνο ζώα προσφαγή ή κτηνοτρόφια, όχι όμως για εκτροφή ταύρων για ταυρομαχίες. Η κτηνοτροφη οχι ομως για εκτροφη ταυρων για ταυρομαχιες η κυρια Μα... Μαρτίνες μίλησε για το γεωρικό εισόδημα και τη σχετική ρυθμίση του 2004 Μπορεί να είχαμε αρνητικά αποτελέσματα στα δημητριακά ή στο ελαιόλαδο, αλλά η προστασία των γεωργών γίνεται με πολλά και διάφορα μέτρα. Ο Ισπανικός νόμος είναι μία πτυχή αυτής της προστασίας. Έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική που εξασφαλίζει άλλα επίπεδα προστασίας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη στήριξη προς τους γεωργούς. Επαναλαμβάνω και πάλι τη διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση 47 επιπλέον δισεκατομμυρίων στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Και μην ξεχνάτε ότι το 2013 η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εξασφαλίζει η βιωσιμότητα όλων των παραγωγών σε όλες τις περιφέρειες της Ισπανίας. Έχει μεγάλο παραγωγικό πλούτο η Ισπανία και εξασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα στρατά του σε κάθε άκρη της Ισπανικής επικράτειας. Εκτός από την κοινή γεωρική πολιτική, εφαρμόσαμε και στην Ισπανία μια πολιτική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που απέφερε καρπούς. Ο κύριος Καπούτο μίλησε για το λίγο χρόνο που έχουμε. Όντως, μας λείπει χρόνος για να αποτιμήσουμε καλύτερα τον νόμο σε ό,τι αφορά την ποιότητα έχουμε πρόσφατα θεσπίσει ένα νόμο για τη βελτίωση της ε, ποιότητας των τροφίμων και την εφαρμογή ελέγχων. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερα χένια και στους καταναλωτές, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας προστασία των εμπορικών τελεστών. Δεν παρουσιάσαμε κύριε Πρόεδρε τον νόμο μας στο Συμβούλιο Υπουργών, το κάναμε όμως ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώσαμε την προθυμία μας να διαβιβάσουμε το νόμο για την εύρυθμη λειτουργία της επιστηστικής αλυσίδας στα κράτη-μέλη που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Αλλά επίσημη παρουσία στο Συμβούλιο Υπουργών δεν έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ευρύτατο και δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, επανειλημμένως το εξετάσαμε. Σε λίγο θα ψηφίσουμε και την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Μαγκίνες για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Περιμένουμε και το υλικό που μας υποσχεθήκατε. Γιατί η δική σας τεχνογνωσία και η δική σας εμπειρία θα είναι χρήσιμη και για τις δικές μας εργασίες και ίσως εμπνεύσει και άλλα κράτη-μέλη. Θα αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε την ισπανική εμπειρία και τα ισπανικά μέτρα. Σας ευχαριστούμε, σας συγχαίρουμε και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε αντίστοιχα και πανευρωπαϊκά μέτρα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και για τις κυρώσεις. Σας ευχαριστούμε και θα περάσουμε στο επόμενο μας σημείο Πάντως, με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι ήδη απέφερε καρπούς η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. γιατί υπάρχουν όντως φαινόμενα μονοπωλίου και συγκέντρωσης, αλλά τέτοια παραδείγματα σαν αυτά της Ισπανίας μας δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή στη συζήτηση και σίγουρα το θέμα αυτό θα συνεχίσει να εξετάζεται σε πολλά επίπεδα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και εκτός. Μία σύντομη διακοπή τεχνικού χαρακτήρα, τρία-τέσσερα λεπτά και άμεση επιστροφή για να συνεχίσουμε γιατί είμαστε ήδη πολύ πίσω στο χρόνο. Ευχαριστώ. Yes, yes, yes, yes, we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny punkt. Ωραία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην ώρα της ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση Μαγκίνες Ήδη έχουμε αναφερθεί στο θέμα. Επιτρέψτε να μου δώσω το λόγο στην εισηγήτη, κύριε Μαγκυρέζα. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να ψηφίσετε. Δύο λόγια για τους κοιόδες εισηγητές. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά ως ομάδα και προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλα τα θέματα στη Συμβαστική Συμφωνία. Καταφέραμε να μειώσουμε, να περάσουμε στις 50 ψήφους. Υπάρχουν ορισμένε ψηφοφορίες που θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ αυτών, αλλά θα ήθελα το μήνυμα να είναι συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνώ. Ε, θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, και με τον εισηγητή Γιάκουβετς. Θα σας κρατήσω ενήμερους σχετικά με τις εξελίξεις για αυτό το θέμα και θα οριστεί και ένας καινούριος εισηγητής για αυτό το θέμα. Εάν υπάρξει καθυστέρηση, δεν ξέρω τι θα συμβεί με αυτό το θέμα και θα έλεγα τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, βοηθό μου, Αλμαρή, την Γραμματεία και τον Άλμο Στρέιτσα για την καθοδήγηση από πλευρά του. Σας ευχαριστώ. Ε, Σίγουρα αν λάβει υπουργικά καθήκοντα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως είπατε. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα λεπτάκι ακόμη. Περιμένουμε τον κύριο Ταραμπέλα να ψηφίσει. Ψηφίσατε. E, Επανάληψη της ψηφοφορίας. Ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 25. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 34. Κατά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 34. Τέλο ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική 5. Πάμε στην τροπολογία 69. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 69. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Καλά που το ελέγξαμε. 59. Τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 59, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 6 τώρα. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. κατά απορρίπτεται μάλλον αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 80 τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 7 τώρα Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 133. Ποιος είναι υπέρ. 133 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για την 133 Zamykam głosowanie. Τέλος. Δεκαοχτώ προς 22 απορρίπτεται. Τροπολογία 127. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Εγκρίνεται. 84. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 131. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 28. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86, Κέστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 105 έρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Odrzucona. Poprawka. Απορρίπτεται. Τροπολογία 163. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 167. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 176. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 177. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 178. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. 180. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 181 άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 184. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 182. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. «182» ηλεκτρονικός έλεγχος για την 182 και πάλι. Τέλος. Εγκρίνεται. 183. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 183. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 185. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 185. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 189. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 189. Τέλος. Με δύο ψήφους διαφορά απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 190 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 191 υπέρ εγκρίνεται 192 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 193 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 146 ποιος είναι υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Τέλος. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Οπότε ψηφίζουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Μαγκίνες. Ξέρουμε τι προβλήματα αντιμετωπίσατε με τις τροπολογίες. Έχετε να προσθέσετε δύο λόγια για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Πολύ σύντομα, σας ευχαριστώ και πάλι. Το ότι ψηφίσαμε προς τη μία κατεύθυνση και όχι την άλλη δεν σημαίνει ότι θα μας στηρίξει και η Ολομέλεια εκτός και αν τονίσουμε τη σημασία της αλυσίδας εφοδιασμού και συνεργαστούμε και με την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ε, παρακαλώ λοιπόν για την συνέχιση της υποστήριξής σας. Ευχαριστώ. Ε, εκ μέρους ε, της Ευρωπαϊκής ε, εκ μέρους της Επιτροπής μάλιστα θέλαμε να απευθύνουμε θερμή έκκληση προς τις πολιτικές ομάδες. Ε, συζητήστε το θέμα αυτό ώστε να μην πάδει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια από αυτό της Επιτροπής. Παρακαλώ καθένα στην ομάδα του να το θέσει για να προλιάνει το έδαφος για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Προχωράμε. Πριν περάσουμε στο σημείο 13, την ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Πιμ Βαμπάκαϊνεν, ο οποίος έχει έρθει και τον καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση, τον κύριο Πιμ Βαμπάλεκο, πρέπει να διεκπαιρεώσουμε το σημείο 12, την ε, εισαγωγή εκτακτών αυτόνομων εμπορικών μέτρων με τη δημοκρατία της Τινησίας. Η συγκήτριά μας εδώ είναι η κυρία Αγγιλέρα που θα συντάξει γνωμοδότηση, ενώ αρμόδια κατ' ουσία είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Παρακαλώ την κυρία Αγγιλέρα να μας παρουσιάσει εν συντομία τη γνωμοδότησή της. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης γιατί εμείς μόνο γνωμοδότηση συντάσσουμε, δεν είμαστε αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή. Πρόκειται για μία πρόταση της Επιτροπής που στόχο έχει την εισαγωγή έκτακτων εμπορικών μέτρων για την, την Ισία ε, για να διορθωθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ιουνίου και γι' αυτό προτείνεται η χορήγηση προσωρινής ε, και μονομερούς δεσμολογικής ποσόστοσης μηδενικού δασμού 35.000 τόνων για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Τινησίας. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, ανησυχία μου πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα για την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συστηματικά Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούν την γεωρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευνοήσουν την διεθνή τους πολιτική. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την προσφυγική κρίση, για παράδειγμα. Και θα ήθελα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στην διαχείριση και τη μετώπιση της προσφυγικής χρήσης. Αλλά να μην χρησιμοποιούμε τη γεωργία ως αντάλλαγμα για να πετύχουμε χάρες ή να κάνουμε χάρες προς μια χώρα. Δεν είναι διαπραγματευτικό εργαλείο η γεωργική πολιτική. Γιατί ήδη ε, η Τινησία δικαιούται ετησίω ποσόστοση 56.700 τόνων ελαιολάδου. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, στο παρελθόν δεν κατάφερε να εξαντλήσει αυτή την ποσόστοση η Τινησία. Και στην ε, νέα πρόταση προτείνεται αύξηση κατά 35.000 τόνους ετησίω για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Τινησίας για να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο ο κλάδος. Η, η τη της έκθεσης ε, έχει τη δική της θέση ε, και εγώ συμφωνώ με την αρχική πρόθεση να βοηθήσουμε την Τινησία για να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα, ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική επίθεση. Αλλά εγώ επειδή κατάγομαι από μια περιοχή που έχει παραγωγή ελαιολάδου και μάλιστα στην Ανδαλουσία 300 κοινότητες και χωριά εξαρτώνται από την εκμετάλλευση των ελαιοδέντρων και την παραγωγή ελαιολάδου Είμαι κατά της αύξησης αυτής της ποσόστοσης ε, κατά 35.000 τόνους για την Τινησία, πολλό δε μάλλον που η Τινησία μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να εξαντλήσει την ποσόστοση που ήδη δικαιούται, χωρίς την επέκταση. Και παραλαμβάνω, δεν θέλω να χρησιμοποιείται η γεωργία ως ε, ε, αντάλλαγμα σε διαπραγματεύσεις άλλης φύσεως. Θα ήθελα με την γνωμοδότηση αυτή να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς την Τινησία, εννοείται, υπό όρους όμως και υπό προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να θέσουμε κάποιους όρους, γιατί είναι σημαντικό και για τη Γενική Πολιτική Συμφωνιών Σύνδεσης και για την ε, συνηθισμένη χρήση που κάνουμε στη διεθνή πολιτική των ε, γεωργικών ανταλλαγμάτων που δίδουμε. Δεν θα πρέπει ο γεωρικός μας κλάδος να πληγεί από αυτή την αύξηση της ποσόστοσης και από τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργείται μερικές φορές εξαιτία των συμφωνιών σύνδεσης. Λέμε ναι στη διαπραγμάτευση, αλλά όχι ανεφόρον. Ναι υπό όρους. Και σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ με αύξηση και προσωρινή ε, δασμολογική ποσόστοση. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτες επιπτώσεων τέτοιων μέτρων στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γιατί αν αυξήσουμε την ποσόστοση ή θεσπίσουμε νέα ποσόστοση, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε κάνει μελέτη επιπτώσεων αυτού του μέτρου στις ε, περιφέρειες. Γιατί θεωρώ ότι στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, στις μεσογειακές χώρες τι συνέπειες θα έχει αυτή η αύξηση της ποσόστοσης ελαιολάδου προς την Τινησία. Και δεν μιλώ μόνο για αυτή την ποσόστοση, μιλώ και για άλλες περιπτώσεις. Γιατί δεν έχει γίνει προηγούμενη μελέτη επιπτώσεων πριν προταθεί αυτό το μέτρο. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι όντως έκτακτα. Έκτακτα και κατεπήγοντα. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την διετία ή να αναθεωρούνται και να παρατείνονται. Επαναλαμβάνω, μέτρα εκτάκτου ανάγκης, κατεπήγοντα και έκτακτα, χωρίς παράταση και επίσης να ε, μην ε, ζητούμε αιτήσια πιστοποιητικά. Γιατί αυτά τα αιτήσια πιστοποιητικά δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσουν περισσότερα ε, τα, τους καταναλωτούς παραγωγούς. Προτιμούμε τα μηνιαία πιστοποιητικά. Μηνιαία πιστοποιητικά οπωσδήποτε, όπως έχει μέχρι τώρα για να παρακολουθήσουμε καλύτερα την επίπτωση. Επίσης, ε, αν εγκριθεί η αύξηση της ποσότητας για την, την, Ισία, θα έχουμε τελικά 91.700 τόνους ίδια ποσόστοση με της Πορτογαλίας που είναι ευρωπαϊκή χώρα. Προσοχή λοιπόν. Αυτή η απόφαση θα επηρεάσει ιδιαίτερα κάποιες περιφέρειες όπως την Ανταλουσία. Και ναι μεν θέλουμε να βοηθήσουμε την Τινησία, θέλουμε να τη συμπαρασταθούμε, αλλά προσοχή. Προσοχή μην πλήξουμε έτσι ανεπανόρθωτα τον κλάδο του ελαιολάδου στην Ισπανία και στην Ανταλουσία. Ευχαριστώ κύριο Δεκάστρο. Θα ήθελα πραγματικά να υποστηρίξω τη γνωμοδότηση της Αντιπροέδρου Αγγιλέρα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα να έχω την προσοχή όλης της Επιτροπής. Συμφωνούμε απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη κρίση που πλήττει την Τινησία. Αλλά δεν μπορούν όλα να φορτωθούν στη Γεωργία και δεν μπορούμε να φορτώσουμε όλα αυτά μόνο σε ένα τομέα της ε, ε, ε, Γεωργίας. Ε, με το θέμα αυτό, ασχοληθήκαμε σε αυτή την Επιτροπή. Ξέρουμε ότι η χρονιά αυτή ήταν ιδιάζουσα, αντιμετωπίστηκαν ξεχωριστές δυσκολίες και εμεί αυξάνουμε τις ποσοστώσεις για δύο χρόνια με ένα ποσοστό που είναι το 20-30% της εθνικής παραγωγής της Ιταλίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό παραμένει βεβαίως το γεγονός ότι σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την Τινησία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όσοι ζητήσουν το λόγο να μην ξεπεράσουν το ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ πολύ την πρόταση της Επιτροπής. Ήταν ένα μέτρο περιορισμένο χρονικά για να εφαρμοστεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην ε, την και θα είχε μία ε, περιορισμένη επίπτωση σε χρόνο. Θα αφορούσε λοιπόν ε, και ο αδασμολόγητης ποσοστός. Νομίζω ότι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ιδιαίτερα γιατί είναι τόσο σημαντικό για την, την, για την οικονομία της ε, την Ισίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να υποστηρίξω την παρουσίαση της κυρίας Αντιπροέδρου Αγγιλέρα. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικά τα όσα είπε. Η Τινησία διανύει σε μια σημαντική ιστορική στιγμή. Πιστεύω ότι το κατεξαίρεση αυτό μέτρο θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι σημαντικό. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει και αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν. Αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στην κατάσταση. Ε, Ο uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα θέλαμε να στηρίξουμε και ενδιαφέρει και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έλεγα λοιπόν ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Θα πρέπει να μην είμαστε τοπιστέ και πραγματικά πρόκειται για ένα τεχνικό ντοσιέ, για ένα ιδιαίτερα πολιτικό θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι αυτό είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να τεθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που αφορά την ε, ε, νότια γειτονία δεν είναι δεδομένη η ιδέα ότι θα μπορεί να υπάρξει δημοκρατική πρόοδος ε, στην ε, την Είναι πολύ πιθανόν η την να βρεθεί αντιμέτωπη με μία σειρά από προβλήματα και θα πρέπει να μας απασχολήσει η οικονομική ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα και στις και υγείας χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ανασκόπηση της πολιτικής μας. Θα υποβάλω αυτή την πρόταση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συζήτηση καθώς και μια κοινή για να δούμε πώς η Γεωργία θα μπορούσε να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Όπως είπαν ε, οι συνάδελφοι, αυτό το μέτρο περιορίζεται χρονικά και εμάς μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Ευχαριστώ κυρία Εράς Γκαρσία. Εγώ είμαι κάθετη και κατηγορηματικά αντίθετη ε, κατά της τρομοκρατίας και σίγουρα είμαι στο πλευρό του λαού της Τινησίας ε, και συμπαρίσταμαι και είμαι υπέρ της γενοδορίας ε, προς τη χώρα αυτή και φυσικά θα πρέπει να την χείρα βοηθείας. Πρόκειται όμως για μία συγκυρία και θα πρέπει αυτό το συγκυριακό χαρακτήρα να έχει και το μέτρο και να είναι προσωρινό και εφήμερο. Δέχομαι την πρόταση ε, του Συμβουλίου και της κυρίας Μογκερίνη αλλά να τροποποιήσουμε κάπως την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκήτρια μας παρουσίασε με πολύ σαφήνεια ε, την κατάσταση. Και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κιλέρα, τη συντάκτρια της γνωμοδότησής μας. Γι' αυτό και θα προτείνουμε μια αλλαγή στο σημείο 9. Το έκανε και η συγκήτρια εγώ θα αλλάξω περισσότερα την τροπολογία της ηγετρίας και θα ήθελα να προσθέσω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί προηγούμενο ε, για την ε, συμφωνία σύνδεσής μας με την Τινησία. Γιατί προς το παρόν είναι άγνωστες οι επιπτώσεις αυτού του μέτρου το 2017 και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την συντάκτρια της γνωμοδότησης που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπε, ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της εισηγήτριας ως προς την ανάγκη του να βοηθηθεί ο, ο λαός της Ισία. Αυτό δεν μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις όμως σε έναν και μόνο τομέα της Γεωργίας. Και συμφωνώ απόλυτα ε, και με τα όσα ανέφερε η εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την κατεξαίρεση φύση και τον περιορισμένο χαρακτήρα της παρέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχεται διαρκώς η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Βεβαίως αυτή η ποσόστοση δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση στις εισαγωγές, θα μπορούσε όμως να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επηρεάσουμε περισσότερο τα πράγματα και να ε, υπάρξει μεγαλύτερη εξέταση, ε, περαιτέρω εξέταση του θέματος από πλευρά της Επιτροπής. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε, θα πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε με αυτή την ε, συμφωνία. Στόχος μας είναι να επιδείξουμε αλληλεγγύη σε μια γειτονική χώρα. Είναι αλήθεια ότι η Γεωργία αποτελεί φορέα πολλές φορές αυτού του είδους ε, της αλληλεγγύης οι 35.000 ε, τόνοι είναι ένα μέρος της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη, θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Ελπίζουμε τα μέτρα που προτείνει η να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενδεχομένως είναι πολύ απαιτητικά, παρόλα αυτά χαίρομαι ε, που έχουμε τη δυνατότητα να εκφέρουμε την άποψή μας. Η γνωμοδότηση της Γεωργικής Επιτροπής είναι θετική στις δύσκολες στιγμές αυτές που διανύει η, την Ισία και στις προσπάθειες που καταβάλει για να βρει μια διέξοδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοιτάξτε, εμένα δεν με χαροποιούν είναι αυτά τα μέτρα. Πιστεύω ότι στρέφονται κατά των ε, γεωργών η κατάσταση στην Ισία οδήγησε σε ένα πολιτικό αντιέξοδο και σε μια κρίση για την οικονομία. Ε, σήμερα μας ζητάνε να ευνοήσουμε την γεωργική παραγωγή ελαιολάδου στην Τινησία, στην εσωτερική αγορά. Όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας σημαίνει ότι ζητάμε από τους γεωργιούς γούρβας να θυσιάσουν έναν ακόμα τομέα της γεωργίας, τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, για να χρηματοδοτήσουμε ένα διπλωματικό φιάσκο. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που είναι κατεπήγον για μας είναι καλά, καταρχάς να εξετάσουμε την κατάσταση των ελαιοπαραγωγών στην Ιταλία και την Κωσική. Το αίτημα που υποβάλλεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι είναι μια καινούρια μαχαιριά. Γνωρίζουμε τις ε, δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γεωργοί και δεν, δεν θα λέγω ότι με πλήση η άποψη των συναδέλφων από την Ευρώπη που σήμερα δεν υπεραμείνονται του πλούτου της περιοχής τους. Πιστεύω ότι θυσιάζουμε ακόμα ένα μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας στο βωμό πολιτικών παιχνιδιών. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη διάταξη γιατί 70.000 τόνοι ε, είναι μια ζημία, μια ζημία για την οικονομία. Βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε την, το λαό της ισία, αλλά όχι με αυτό το τίμημα. Αυτό είναι μια ζημία για την οικονομία, το χωρό της Νότιας Ευρώς, για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Νότια Ιταλία. Ενώ ε, αυτοί στην ε, Βόρειο Ευρώπη δεν θα τηγούν που δεν είμαι αυτό το μέτρο. Και πάλι συνεπώς πλήττουμε χώρες οι οποίες διανύουν μια προβληματική περίοδο, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας. Αυτό είναι ένα μέτρο που δεν μας βρίσκει σύμφωνους γιατί υπάρχουν και άλλοι μέσα μέσω του προγράμματος μικροοικονομικής βοήθειας το 2011 δόθηκαν 800 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα διοχετεύτηκαν 100 εκατομμύρια το η πρώτη δόση μιας ενίσχυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι μια ε, ένα μέτρο που δεν μας βρίσκει σύμφωνους, κυρίως ε, όταν ε, ανακαλύπτουμε ότι μεταξύ των μεγαλοπαραγωγών ελαιολάδου είναι ο Πρωθυπουργός της Τινησίας. Στην ουσία ξεπουλάμε την γεωργία σε αντάλλαγμα πολιτικών παιχνιδιών. Το κάναμε με τα εσπεριδοδοί στο Μαρόκο, με το ρύζι στην Ασία και τώρα το ξανακάνουμε την Τινησία και το ελαιόλαδο. Ευχαριστώ. Και τώρα η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η κυρία Σπυρός, παρακαλώ, έχει το λόγο. Good morning. Ε, Καλημέρα. Ε, ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες καταγωγής, η Κομισιόν στηρίζει την τροπολογία, η νέα διατύπωση ευθυγραμμίζεται και με τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης σχετικά με την υποχρέωση για μελέτη επιπτώσεων θυμίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν ελήφθη μετά από μια έκτακτη κατάσταση στην Τινησία και επειδή είναι επίγουσα η κατάσταση δεν μπόρεσε να γίνει μελέτη επιπτώσεων, μελέτη αντικτύπου. Όμως η Κομισιόν ανάλυσε την κατάσταση της αγοράς και θεωρεί ότι το μέτρο δεν θα πλήξει αρνητικά τους ε, παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κάτω λόγους. 35.000 τόνοι αύξηση είναι μόνο 2,2% ε, της κατανάλωσης του 2014 και του 2015 στην Ένωση. Η το ελαιόλαδο και τα αποθέματα ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ε, στο τέλος της ε, περίοδου 11-12 τα αποθέματα ήταν 887.700 τόνοι, ενώ τώρα εκτιμώνται σε 317.400 τόνους και δείκτες δείχνουν ότι η ενωσιακή παραγωγή για την επόμενη περίοδο, 15-16 δηλαδή, δεν θα είναι επαρκώς σημαντική ώστε τα αποθέματα της Ένωσης να φτάσουν στον ιστορικό μέσο όρο τους. Επίσης, λόγω της χαμηλής παραγωγής του προηγουμένου έτους εμπορίας, οι ντόπιε τιμές, οι εγχώριες τιμές είναι σε χαμηλό ρεκόρ και ήδη άρχισαν οι εισαγωγές ε, ελαιολάδου από την Τινησία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Έτσι, ο κίνδυνος είναι η τωρινή αύξηση τιμών ελαιολάδου να οδηγήσει τους καταναλωτές και τη βιομηχανία τροφίμων να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά προϊόντα μέσω και μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει τους του συνεγγύς εισαγωγές ελαιολάδου ε, στα πλαίσια των δεσμολογικών ποσοστώσεων νέων και τρεχουσών για να δει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές του ελαιολάδου και θα εξετάσει αν χρειαστεί προτάσεις για τα κράτη-μέλη αν υπάρξουν σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά ελαιολάδου. Δεν χρειάζεται να δοθεί ε, η αρμοδιότη στην Επιτροπή να προχωρήσει σε προτιμησιακή συμφωνία. Ο ο κανονισμός 1408 ε, δίνει ήδη εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις, ιδιαίτερα ε, αν ε, χρειαστούν ε, διαφοροποίηση. Εις ό,τι αφορά το θέμα των πιστοποιητικών εισαγωγή, η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση εδώ, διότι δεν θα επηρεάσει τις εισαγωγέ του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, επειδή η άδεια που δόθηκε τέλος Οκτωβρίου θα ισχύει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Για λόγους απλούστευσης και διευκρινήσεων, η διαχείριση των αυτόνομων ποσοστώσεων και των ε, ε, δασμολογικών ποσοστώσεων θα πρέπει να είναι παρόμοια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ε, κυρία Αγγιλέρα, αλλά σας θέλω παρακαλώ ένα λεπτάκι μόνο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Τους ευχαριστώ για τις προτάσεις τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες και σύντομα να ψηφίσουμε κιόλα. Η Επιτροπή η Διεθνούς Εμπορίου είναι αρμόδια κατ' ουσία Επιτροπή που στην αρχή μας ε, ζόρισαν προκειμένου να διεκπαιρώσουμε πολύ γρήγορα την ε, σύνταξη της γνωμοδότησης και μετά οι ίδιοι παρέτεναν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να παρατείνουμε και το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να πω στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους συναδέλφους το εξής. Όντως, το ελαιόλαδο, η ποσόστοση αυτή επηρεάζει τους παραγωγούς του Νότου. Τη Μεσογείου. Και είμαστε ιδιαίτερα γενναιόδοροι δεδομένης κατάστασης γιατί πραγματικά η Τινησία το αξίζει. Και θα υπερψηφίσουμε αυτό το μέτρο με τις παρατηρήσεις όμως που έκανα και τι επιφυλάξει που σα εξέθεσα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα. Όντως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα για την εσοδιά και την περίοδο 2015-2016. Αν όμως διαπιστωθεί σημαντική διατάραξη της αγοράς ελαιολάδου ε, αργότερα, παρακαλώ να δείξει ευαισθησία και ως προς την ιδιωτική αποθεματοποίηση αργότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 18 Νοεμβρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, 11 το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την ε, υποβολή των τροπολογιών. Θα ε, ψηφίσουμε στην 1η Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και τώρα καλωσορίζω στο βήμα τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕ. Το θέμα της γνωμοδότησης για την γεωργία στις ορεινές περιοχές αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. Οπότε δεν υπάρχουν παρατηρήσεις και για τις συστάσεις των συντονιστών. Θεωρώ ότι εγκρίνονται οι συστάσεις των συντονιστών. Έχετε λάβει τις συστάσεις και γραπτός, οπότε τις εγκρίνουμε και καλωσορίζουμε θερμότατα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Πιμ Βαν Μπάλεκομ. Τον Αύγουστο, ο κύριος Βίλι Μόρτερ αποχώρησε από την ΕΤΕ και το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας ανέλαβε ο αντιπρόεδρος απίν Βαμπάλεκομ πριν από ένα μόλις μήνα. Χαιρόμαστε γιατί ήδη είναι δυνατή πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕ που είναι σημαντικότατος εταίρος στη Γεωργία Έχουμε σημαντικές αλλαγές στο τοπίο το ευρωπαϊκό σε πολλά θέματα και χαιρόμαστε για τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τον Αντιπρόεδρο. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε και περιμένουμε την παρουσίασή σας. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, πριν από λίγους μήνες, την 1η Σεπτεμβρίου, ζήτησα από τον πρόεδρό σας να διοργανώσει μια σύντομη συνάντηση για να σας παρουσιαστώ και είπε καλό θα ήταν αυτό, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να έρθετε για να σας δει όλη η Επιτροπή και όχι μόνο εγώ. Ήρθα λοιπόν χάρη στον πρόεδρο, ο οποίος έκανε την πρόταση. εκλήθη να αναλάβω θέματα αγροτικά στην Τράπεζα Επενδύσεων μετά την αποχώρηση Μόλτερερ και δέχθηκα, όχι μόνο γιατί μου το ζήτησε ο πρόεδρος, που βέβαια αυτό είναι ένα βαρύνον επιχείρημα πάντα, αλλά είχα κίνητρο για να ασχοληθώ με τα τρόφιμα και τη βιομηχανία τροφίμων. Όχι μόνο γιατί προέρχομαι από αγροτική περιοχή και επειδή η μητέρα μου εξακολουθεί να ζει σε αγρόκτημα, όχι βέβαια δραστήρια πια, αλλά είναι 85 ετών, μην το ξεχνάμε, υπάρχει διαφορά ηλικίας της επιτρέπεται να είναι λιγότερο δραστήρια από ό,τι ήταν. Το βασικό μου κίνητρο ήταν ότι ο τομέας της γεωργίας είναι κρίσιμος για μια ανθυρή ευρωπαϊκή οικονομία. Και η αλληλεία, η δασοκομεία, τα τρόφιμα, εκτός από τη γεωργία, αποτελούν βασικούς πυρήνες της ευρωπαϊκής οικονομίας και απασχολούν περίπου 12 εκατομμύρια αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ε, είναι σωστά τα στοιχεία μου, 1,4 εκατομμύρια ε, εταιρείες μη αγροτικές και δίνουν εργασία σε 85 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανταγωνιστική γεωργία σε ένα ανταγωνιστικό τομέα έχει σημασία για, για πολλούς λόγους. Δηλαδή βελτιώνει τη συνοχή στις ε, αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο, είναι σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, γιατί αν η οικονομική ανάπτυξη επανέλθει σε τροχιά καλή στην Ευρώπη, σε κάποιες περιοχές της Ένωσης ή τα ποσοστά ανεργίας είναι παράδεκτα υψηλά και ο τομέας της γεωργίας μπορεί να παίξει κέριο ρόλο εδώ. Είναι καλή η ανάπτυξη εδώ και για τις καινοτομίες και τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Πολλοί τομείς λοιπόν επηρεάζονται από μια ανθυρή γεωργία. Μετά από 20 χρόνια υποεπενδύσεων στην αλυσίδα τροφίμων και στο γεωργικό τομέα σε πολλές ε, χώρες, τώρα χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, ούτω ώστε η υποδομή, η πεπαλαιωμένη, ε, όπως και οι εξοπλισμοί, τα εργαλεία να ε, ανακαινιστούν. Αυτό μπορεί να γίνει νομίζω με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα παράλληλα πάντα με τις πολιτικές της Ένωσης. Και νομίζω ότι ο τομέας ε, γεωργίας και τροφίμων έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Ένας δεύτερος ρόλος ε, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, κλήθη από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να δράσει περισσότερο για η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών εταιριών. Θα γνωρίζετε ότι ένα συμπέρασμα που έγινε πέρσι δεκτό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η προώθηση και η υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιριών ώστε αυτές να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στη διεθνή αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η τράπεζα βεβαίως είναι μια τράπεζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το 90% του όγκου εργασιών μας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 10% του όγκου εργασιών μας λαμβάνει χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, περίπου 8 δις ετησίως είναι αυτό. Είμαστε δραστήριοι, για παράδειγμα, στη Σενεγάλη, παράδειγμα λέω τώρα, και άλλες χώρες ΑΚΕ και νομίζω ότι αυτό καλό είναι να το έχουμε υπόψη. τα τελευταία πέντε χρόνια ε, ε με την, υπό την ηγεσία του καλού μου φίλου Μόλτερερ 20 ε, δις ευρώ ως δάνεια δόθηκαν στη γεωργία, Αλληλία και δασοκομεία και τις, τους συναφείς κλάδους. Και πάντοτε ο Μόλτερ έλεγε και εξακολουθεί να είναι αυτό το μότο της τράπεζας ότι η τράπεζα είναι για να δανειοδοτεί, να αναμειγνύει ε, στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επίσης ε, ε, βοηθούμε μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών τα κράτη-μέλη εκ των προτέρων αναλύσεις για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μια προτεραιότητα είναι βεβαίως η ανάπτυξη ε, προγραμμάτων εγγυήσεων για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στις, στον τομέα των ΜΜΕ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι ο πιο σημαντικός στο, στη γεωργία. Συνεργασία προβλέπεται επίσης και στενή συνεργασία για υποστήριξη της έρευνας και ε, δυνατότητες ε, επίδειξης για πρώτη φορά ε, στα λεγόμενα νέα προϊόντα ε, βεβαίως, θέλω, επειδή εδώ ήρθα για ανταλλαγή απόψεων, θα είμαι σύντομο. Δύο παρατηρήσει θα κάνω ακόμη. Πρώτον, ε, το πρόγραμμα Juncker, το σχέδιο Juncker, νομίζω ότι το μέσο τη Γεωργίας θα ωφεληθεί από τι επενδύσει που είναι γνωστέ στο σχέδιο Juncker. Η Κομισιόν θα δώσει εγγυήσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτω ώστε να αναλάβει ε, μεγαλύτερο κίνδυνο στι επενδύσει. και αυτό μπορεί να ανοίξει νέε δυνατότητε για τον τομέα αλλά και για την τράπεζα. Τώρα αναπτύσσουμε σε αυτά τα πλαίσια νέα προϊόντα όπως εγγύησεις προς τις τράπεζες για χαρτοφυλάκια δανείων προς νέους αγρότες και οι διαδόχους τους ε, ή ε, μεγαλύτερη ε, επένδυση σε μία δασοκομείας, επίσης προγράμματα επιμερισμού του κινδύνου που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη μία πλευρά να αυξήσει τα δάνεια στο τομέα της γεωργίας και από την άλλη πλευρά να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο στις συναλλαγές. Ε, ήδη, έχουν εντοπιστεί νέοι πελάτες εδώ, όπως ε, ε, τράπεζες γέφυρα και άμεση, δα, άμεσος δανεισμός σε γεωργικούς συνεταιρισμούς που είναι ένας νέος τομέας αυτός. Τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε, ως εταιρεία, μια εταιρεία ή ένας τομέας, γιατί θέλει να ε, έρθει σε επαφή και να συνεργαστεί με την Τράπεζα Επενδύσεων. Πρώτον, είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές. Αυτό είναι πάντα καλό, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις. Ε, δεν αναθέτουμε ε, τη, η πολιτική μας δηλαδή δεν είναι crowding out, είναι crowding in δεν ζητούμε κεφάλαια από όλους τους συντελεστές το δεύτερο πλεονέκτημα είναι η ε, μεγαλύτερη διάρκεια ληξιπρόθεσμων δανείων που χορηγούμε, πράγμα που χρειάζεται προκειμένου περί καινοτομιών και επενδύσεων. Η τεχνική μας συμβουλευτική υπηρεσία, από ό,τι λένε όλοι, είναι πάρα πολύ καλή και η διαδικασία δέουσας επιμέλειας για τον εμπορικό τομέα διευκολύνεται έτσι. Έχουμε καλές σχέσεις με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και γνωρίζουμε τους κανόνες λειτουργίας ε, και αυτό ε, δεν το γνωρίζουν πάντα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να ε, παίξουμε ρόλο και να μεσολαβήσουμε, γιατί ξέρουμε τους κανόνες, και η διαφοροποίηση της χρηματοδότησης πάντα είναι καλή για μια επιχείρηση. Και να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας χρηματοοικονομικός εταίρος, ακόμα και σε περιόδους ισχνών αγελάδων για την οικονομία. Ε, είμαστε αντι-αντικυκλικοί. Έτσι το λέμε στην πολιτική μας. Δηλαδή παραμένουμε στην αγορά ακόμα και όταν ο εμπορικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ή δεν του επιτρέπεται να επενδύσει σε τομείς υψηλού ρίσκου λόγω υφισταμένων κανονισμών. Ε, Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή όπου καλείται ο, η, ο εμπορικός τομέας να κάνει απομόχλευση ή να κάνει πίσω. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε απομόχλευση και ζητούμε από τους μετόχους να κάνουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε και υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο γεωργικός τομέας είναι από τους πιο σημαντικούς στην ευρωπαϊκή οικονομία. Προσβλέπω λοιπόν σε μια ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα επόμενα χρόνια αν ε, έχετε ερωτήσεις, ε, ακόμα και στο τέλος της συνεδρίασης αυτής, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου και με τους συνεργάτες μου και είμαι βέβαιος ότι θα ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις σας. Μπορεί να μην, απαντηθούν, να μην απαντώνται πάντα θετικά, αλλά θα απαντηθούν και θα εξηγηθεί σε σας γιατί δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε θετικά αγαπητοί ευρωβουλευτές, ακόμα βρίσκομαι μέσα στην καμπύλη μάθησης. Οπότε μπορείτε να με βομβαρδίσετε με ιδέες, προτάσεις και εγώ θα δω μαζί με τους συνεργάτες στο Λουξεμβούργο να δω αν μπορώ να προσθέσω κάτι στο κλάδο της Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχουν εγγραφεί στο κατάλογο μιλητών Μαγκίνες Δέσσερα, Σένερα και Αγγιλέρα. Χαίτεμα και Καπούτο. Δύο λεπτά καθένας. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Έχω μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν κάνατε αναφορά στην πρόσβαση σε πιστώσεις για τους μεμονωμένους γεωργούς. Θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτό το θέμα. Επιτρόπος Χόγκαν κατά τη διάρκεια των, των καλοκαιρινών μηνών ανέφερε ότι θα μπορούσε να ήταν αυτό μια δυνατότητα. Και πολύ συχνά με ρωτάνε στην Ιρλανδία είναι πότε θα έρθουν τα χρήματα, πώς θα υποβάλω το αίτημα, θα είναι 3%, θα είναι για ένα διάστημα 20 ετών, θα μας ε, βοηθούσε λοιπόν αν θα μπορούσατε να διευκρινίσετε τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε. Ύστερα ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών σε αυτή τη σχέση αν θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε χρηματοδοτήσεις στους γεωργούς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε σκεφτεί κάτι για τους νέους γεωργούς. Εδώ μιλάμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑ, προσπαθούμε να θαρρύνουμε μια νέα γενιά, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη η γενιά αυτή με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τα έσοδα από την γεωργία μπορεί να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα μου ερωτήματα. Ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΤΕ σε ό,τι αφορά την κοινότητα των γεωργών και με μονομένους γεωργούς. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε και διάδοχε του κυρίου Μόλτερ τον ήξερα καλά. Παρουσιάσατε και τα δικά σας θέματα και το πρόγραμμα. Ευχαριστώ που είπατε ότι 25 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τη Γεωργία. Εγώ είμαι από τη Βαβαρία, όπου έχουμε πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αλλά Παλιά ο τομέας αυτός ήταν, είχε την υψηλότερη απασχόληση πιο πολύ και από τον κατασκευαστικό τομέα ε, και τη βιομηχανία. Τώρα, σχετικά με τις προσφορές σας, η κατάσταση στην Ευρώπη διαφοροποιείται βεβαίως. Ε, πρόσφατα ε, ακούσαμε για μια προσφορά στη Raiffeisen ε, σταθερό επιτόκιο 1% για 12 χρόνια, σταθερό επιτόκιο 1,5%. Ε, είναι οι δικές σας ε, προσφορές πιο οικονομικές, γιατί θα μπορούσαμε να το δούμε. δεν ξέρω πώς θα είναι τα επιτόκια μετά από 20 χρόνια ή σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Γιατί το είπα στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Εμείς έχουμε χαμηλά επιτόκια, τόσο χαμηλά που δεν τα ε, έχω ξαναδεί. Και σίγουρα αυτό θα είναι ενδιαφέρον για κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Άλλο ενδιαφέρον που το είπατε ήδη. Σε ποιο βαθμό είναι πρόθυμη η τράπεζά σας να μπει σε κεφάλαια κινδύνου, γιατί αυτό για ορισμένους γεωργούς, το είπατε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ χαίρομαι που θα έχουμε μια καλή συνεργασία και ελπίζω ε, με τη, στην επόμενη ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε για όλα αυτά. Υπάρχουν μερικά ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω στον Αντιπρόεδρο. Ε, επειδή στη Λιθουανία δεν έχουμε πολλούς συνεταιρισμούς ε, και σήμερα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα δήματα ε, αυτών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα υποστηρίξετε τους συνεταιρισμούς στο γεωργικό τομέα. Θα μπορούσατε μήπως να αναφερθείτε σε ορισμένες αρχές πως η δική σας στήριξη στους συνεταιρισμούς θα διαφέρει από τους άλλους. Στη Λιθουανία, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες μένει, πολλά επενδύθηκαν στο γαλακτοκομικό τομέα. Όταν η τιμή ήταν αποδεκτή, ο γαλακτοκομικός τομέας αναπτυσσόταν με γοργούς ρυθμούς. Με την κρίση για δεύτερη χρονιά σαν ε, κράτος αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και οι επενδύσεις είναι μοιραία πάρα πολύ χαμηλές σε αυτό το τομέα. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο το 2% των ε, γεωργών παρετήθηκαν από τον κλάδο αυτό της παραγωγής σταμάτησαν την παραγωγή και προσπαθούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους ξεπουλώντας την περιουσία τους και ο αριθμός των αγελάδων μειώθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον των γαλακτοπαραγωγών στη χώρα μου και γενικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να παίρνουν δάνεια, τα δάνεια που χρειάζονται για ζωτροφές, για βιταμίνες κτλ. Πραγματικά λοιπόν θα με ενδιέφερε να μου πείτε πώς αυτός ο γαλακτοκομικός τομέας καθώς και άλλοι τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για το μέλλον της γεωργίας, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε την διασφάλιση ότι οι τομείς αυτοί θα μπορέσουν να προχωρήσουν και ότι θα, είναι, ε, θα αποφέρουν κέρδη. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση προς τον ε, Αντιπρόεδρο της ΕΤΕ. Όταν μιλήσατε για ε, ενέργειες κινδύνου, τι ακριβώς εννοείτε. Κάποιες συναλλαγές ε, κινδύνου. Η κυρία Αγγιλέρα, ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του Αντιπρόεδρου της ΕΤΕ μας φέρνει πιο κοντά στις δυνατότητες που έχει ΕΤΕ να βοηθήσει τους γεωργούς και τον αγοροεπιστήστικο κλάδο γενικώ, γιατί δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με το έργο της ΕΤΕ οι γεωργοί μας. Συνήθως, όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, ε, οι σχέσεις των Ισπανών με την ΕΤΕ ήταν ε, αιτήσει ε, συνδρομής προς τη διοίκηση. Υπάρχει δυνατότητα παροχής άμεσης συνδρομής προς τους γεωργούς και αν ναι ποιο τρόπο. Αναφερθήκατε στους νέους γεωργούς. Τι δυνατότητες υπάρχουν για να στηρίξετε οικονομικά ή να συμπεριλάβετε και τους νέους γεωργούς στο έργο σας. Πώς μπορούμε να εντάξουμε νέους γεωργούς ε, στους συνεταιρισμούς. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Κύριος Χαϊτεμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε που σκεφτήκατε την Επιτροπή μας. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η εμπλοκή σας. Αναφερθήκατε σε διαφορετικούς ρόλους της ΕΤΕ και τον αγγελικό τομέα. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες γι' αυτό. Πιστεύω, αναφέρουμε σε τρία πράγματα, όπως ανέφερε η κυρία Μαγκίνες, μια καλύτερη πρόσβαση στις πιστώσεις, ιδιαίτερα για τους νέους ε, γεωργούς που θέλουν να αναλάβουν ένα αγρόκτημα. Είναι μια, ε, ένας κλάδος εντατικός κεφαλαίου, συνεπώς είναι πολύ καλό να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης είναι ενδιαφέρον για την ΕΤΕ να σκεφτεί την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών μέσων Ε, ε, ε, θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως οι κακές καιρικέ συνθήκες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ενδιαφέρον αυτό. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει καθ' ολοκληρία από την κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένω σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τρίτον, θα ήθελα να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενδιαφέρεται να επενδύσει σε νέο, νέα πιλωτικά προγράμματα ή νέα ερευνητικά προγράμματα στον κλάδο των μειών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα τα όσα είπε ο κύριος ε, Βαν Μπάλεκόμα. Καταλαβαίνω ότι έχει ένα μεγάλο άνοιγμα λόγω της καταγωγής του προς την ε, Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη έχει αναπτύξει ε, δραστηριότητες στην Ιταλία. Για παράδειγμα, στήριξε πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους, μικρός, ε, και τους νέους γεωργούς. Κάνατε αναφορά στην ε, δράση, την αντικυκλική δράση της ε, ΕΤΕ σε σχέση με τις άλλες τράπεζες. Θα ήθελα να καταλάβω τι είδους πρωτοβουλίες σκοπεύετε να πάρετε σε ένα κλάδο όπως αυτόν της Γεωργίας που χαρακτηρίζεται από όχι υψηλές ε, ε, υψηλά εισοδήματα και όπου ο επιχειρηματικός κίνδυνος έχει σχέση και με εξωγενείς παράγοντες. Οι τράπεζες δεν κινήθηκαν ε, παράλληλα με τον γεωργικό τομέα πάντοτε. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια, ένας διάβλος για αυτόν τον, τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει και συμφωνώ με τον συνάδελφο που πήρε το λόγο πριν από μένα και από την άποψη των ε, εγγυήσεων για ε, να μπορέσει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί κάποιο μέτρο που θα πρόβλεπε, για παράδειγμα, τη δημιουργία ενός ταμείου εγγύσεων που θα επέτρεπε να αντιμετωπιστούν ακραίες καταστάσεις που εμφανίζονται στον κλάδο. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε. Μια συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με την ερώτηση για τα κεφάλαια κινδύνου. Στο γαλακτοκομικό τομέα έχουμε μεγάλη κρίση τιμών. Συζητούμε με τους Ευρωπαίους ε, αγρότες και λέμε ότι μέσω της αποθεματοποίησης και δεν μπορεί η Ευρώπη να καλύψει όλα τα προβλήματα. Δηλαδή ενθαρρύνουμε τους γεωργούς να αναλάβουν δράση και να ρυθμίσουν οι ίδιοι την αγορά και να ε, ε, ε υιοθετήσουν μια αντικυκλική στάση. Βεβαίως ε, όλα αυτά δεν αποδίδουν. Θα πρέπει να δούμε παράλληλα και προγράμματα των συνεταιρισμών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναλάβουν κάποιο ρίσκο αλλά ε, η κρίση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει όρια. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι το νερό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργία και η χρηματοδότηση ε, έργων υποδομών για την άρδευση είναι σημαντικό για τους είναι σημαντικά μέτρα και πρωτοβουλίες για τους Γιώργους. Τώρα, για τους συνεταιρισμού. Αν θέλουν να ξεφύγουν από τις επιχορηγήσεις και τις ενισχύσεις, πώς μπορούν να υποφεληθούν από τα γράμματα της ΕΤΕ. Η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη έχει και ένα στοιχείο κινδύνου. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά τα θέματα και περιμένουμε σε 10 λεπτά να μας διαφωτίσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις μας μου δίνουν την δυνατότητα να εξηγήσω καλύτερα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καταρχάς, και αυτό δεν έχει σχέση με την, τα ερωτήματά σας, από το ξεκίνημα της κρίσης το 2007, η τράπεζα είναι εντελώς διαφορετικός θεσμό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν ήταν, ήμασταν μια τράπεζα υποδομών, η οποία ασχολείται με αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και οτιδήποτε. Βεβαίως, αρτήσουμε δραστηριότητες ακόμα σε αυτό το τομέα αλλά αυτό δεν αφορά το 75% του χαρτοφυλακίου μας, αλλά μόνο το 1-3%. Υπήρξε λοιπόν μία μετατόπιση, μετακίνηση, μία αλλαγή στο χαρακτήρα. Το 1 τρίτο, ως προς το 1 τρίτο ασχολούμεθα με τις υποδονεμές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί ε, αυτό είναι κάτι που πάντοτε χρειάζεται ανανέωση, κατασκευή, συντήρηση υποδομών υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα συντήρησης. Το άλλο, το 1 τρίτο είναι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση όχι μόνο για το γεωργικό τομέα αλλά και για αρκετούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες περιορίστηκε σαν αποτέλεσμα της κρίσης και εκεί ακριβώς δραστηριοποιηθήκαμε και εμείς και το 1 τρίτο είναι ένα κράμα ε, κοινωνικών κατοικιών, ε, κλάδου υγείας, εκπαίδευση κτλ. Άλλαξε λοιπόν ο προσανατορισμός της τράπεζας. Ελπίζω ότι στις ε, επαφές σας με τις ε, συνεταιρισμούς ή με μονομένα άτομα στις χώρες σας θα το πείτε ότι η ΕΤΕ θα μπορούσε να συνδράμει διάφορους τομείς. Δεν είναι μόνο τράπεζα υποδομών. Ε, ταξιδεύουμε βέβαια στην ε, Ευρώπη και πιστεύουμε αν θέλετε το πιστεύετε, έρχονται πολλοί συνεταιρισμοί στην ΕΤΕ που στο παρελθόν δεν θα σκεφτόντουσαν ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει η ΕΤΕ. Τώρα να περάσουμε στα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα ε, από την κυρία Μαγκίνες. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση ε, ε, από, τους, από τον των γεωργών στο παρελθόν στην τράπεζα χρησιμοποιούσαμε τον όρο Hogan Fund, ταμείο Hogan. Μετά τη συνάντηση με την Επιτροπή σας, το συζήτησα, έχω μια συζήτηση με τον Επίτροπο Hogan στη μία, γιατί πραγματικά ασκεί πιέση στην τράπεζα να επιταχύνει κάπως τη διαδικασία αξιολόγησης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά επιταχύνουμε τη διαδικασία.

Βεβαίως, ο εμπορικός τομέας αμέσως λέει ότι θα ε, ε, προτίθεται να το κάνει ο ίδιος. Τη στιγμή λοιπόν που περνάει κανείς στην αγορά, οι άλλοι λένε «Κοιτάξτε, είναι ε, δικό μας θέμα, μην παρεμβαίνετε». Εμείς ως δημόσια τράπεζα θα πρέπει να κινηθούμε σε ένα επίπεδο αν μπορεί να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας, ε, κανένα πρόβλημα. Αλλά το ερώτημά μας είναι γιατί δεν το κάνατε ε, πριν, ε, πριν να γίνουν οι συζητήσεις με τον Επίτροπο Χόγαν, όλα αυτά σε ό,τι αφορά το Γαλακτοκομικό Ταμείο. Υπάρχει λοιπόν το θέμα και θα δούμε τι θα μπορούσε να γίνει. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό θα εφαρμοστεί και ελπίζω ότι θα γίνει με τον ιδιωτικό τομέα. ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος, ε, ένα μεγάλο ίδρυμα, ε, δεν ξέρουμε τις τοπικές αγορές. Στην Γαλλία συνεργαζόμαστε στο γεωργικό τομέα με το κρεντή αγρικό, στην Ολλανδία με, μια, με την Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεργάτε. Υπάρχει όμως η πρωτοβουλία και ο επίτροπο ζητάει από την τράπεζα να επιταχύνει την όλη διαδικασία και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ικανοποιήσω αυτή την επιθυμία του. Ξεκινάμε με ένα Ιρλανδικό γαλακτοκομικό ταμείο και όπως είπε ήδη ο η ιδέα είναι στην Ευρώπη να παρεύουμε εκεί που το ζητάει η αγορά. Εάν υπάρχει δυνατότητα, τότε και αν υπάρχει ένα πλαίσιο μπορεί να αντιγραφεί επακριβώς και σε άλλες χώρες. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που μας απασχολεί ιδιαίτερα τώρα τελευταία. Δεύτερο θέμα. Μας απασχολεί η δημιουργία ενός μέσου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των νέων γεωργών που επιθυμούν να αναλάβουν ε, ε, γεωργικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι εντελώ καινούριο κλάδο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύω όμω ότι αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τι ιδέε του κυρίου Γιούγκερ, θα μπορούσαμε ε, να, να προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε νέα προϊόντα στην αγορά. Νομίζω ότι η κυρία Μαγκίνες μίλησε για τη μεταρρύθμιση, τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτά είναι θέματα που αφορούν τις χώρες μέλη και όχι την ΕΤΕ. Ο κύριος Ντες αναφέρθηκε στο 1,5% σε 112 χρόνια και το ερώτημά του είναι κατά πόσο είμαστε φτηνότεροι. Εκεί βρίσκεται η διαφορά σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από 7 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια η, κράση, η κρίση στην Ευρώπη ήταν μια κρίση ρευστότητας, δεν υπήρχε πρόσβαση στο ρευστό. Τώρα ε, δεν συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Ντράγκη κατακλίζει την Ευρώπη με χρήματα. Παρόλο που τα, τα χρήματα είναι φτηνά, οι επενδύσει δεν προχωρούν με γοργού ρυθμού. Είναι θέμα ανάληψη κινδύνων και όχι τιμών. Η δυνατότητα ανάληψη κινδύνων τη Ευρωπαϊκή οικονομίας συνεχίζει να παραμένει χαμηλή. Γι' αυτό το λόγο είτε την κατάλληλη στιγμή το πρόγραμμα Juncker, γιατί αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει οι τράπεζες να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους και πιστεύω ότι αυτό είναι ο δρόμος για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες, ο κύριο Χάιτεμ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Βεβαίως και ασχολούμεθα και με τις καινοτομίε και ασχοληθήκαμε με τις καινοτομίε και πριν εμφανιστεί το πρόγραμμα Juncker. Αυτό έγινε στα πλαίσια του προγράμματος ε, Horizon 2020 και συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμεθα εδώ. Ελπίζουμε και αναμένουμε να υπάρξουν περισσότερες τέτοιες δράσεις στο μέλλον λόγω του ότι τράπεζα, ε, επιτρέπεται στην τράπεζα να το κάνει αυτό, τη επιτρέπουν οι ε, μέτοχοί της. Και έγινε μια αναφορά στο, και στο εταιρικό κεφάλαιο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι δεν είμαστε μόνο μια τράπεζα δανεισμού ή συμβουλευτικής ή ένας μικτός φορέας. Υπάρχει και ένας κλάδος που αφορά τα ε, κεφάλαια κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Τμήμα Επενδύσεων και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε μη τραπεζική χρηματοδότηση, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται πάρα πολύ στις τραπε... Ε, από την τραπεζική χρηματοδότηση αν λοιπόν έχετε ιδέες οι πελάτες οι συνεταιρισμούς που αναζητούν χρηματοδότηση εκτός τραπεζών, παρακαλώ προωθήστε τους στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να τους φέρουμε σε επαφή με άτομα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που τίθενται πάντοτε ότι την τράπεζα την αφορούν τα μεγάλα ποσά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εμείς κινούμεθα στον ε, εμπορικό τομέα, στις χώρες όπου αναπτύσσουμε δραστηριότητες και ε, ακόμα και σε μικρή κλίμακα μπορεί να γίνει άμεσος και έμεσος δανεισμός ξεκινώντας από τα 5 εκατομμύρια. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για ένα έτος. Μπορεί να κατανεμηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας. Το... Η τελευταία ερώτηση, πληρώ να κατάφερα να απαντήσω σε όλες, αν όχι, σας ζητώ συγγνώμη. Ο πρόεδρος έφυγε, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο πρώτος λοιπόν με ρώτησε αν, αν αναπτύσσουμε δραστηριότητες στον τομέα των υδάτων. Ε, πρόσβαση στο, στο καθαρό είδωρο, πελάτης Βασινιάκου Αφίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον γεωργικό τομέα. Αυτό ισχύει και για τις ε, χώρες για τις οποίες είμαι υπεύθυνο για την υποσαχάρια ας πούμε Αφρική. Εκεί καλούμεθα να κάνουμε περισσότερα στο γεωργικό τομέα. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι παρακείμενες επενδύσεις ε, που απαιτούνται ε, γιατί αν παράγει κανείς και δεν μπορεί να μεταφέρει δεν θα συμβεί τίποτα. Η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι κάτι που ήδη κάνουμε εδώ και αρκετό χρόνο. Εγώ αναφέρθηκα μόνο στα θέματα που μας επιτρέπουν να, προχωρήσουμε περισσότερο στο μέλλον χάρη στο πρόγραμμα ε, Juncker. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, ε, ανάληψη κινδύνων, περισσότερα προϊόντα για τους νέους γεωργούς, περισσότερες κοινοτομίες, ε, διευκόλυνση νέων γεωργών να αναλάβουν τις επιχειρήσεις των γονιών τους ή δημιουργία ενός μηχανισμού με τις εμπορικές τράπεζες για τον γαλακτοκομικό τομέα. Ελπίζω να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στη συνάντηση που θα έχω στη μία με τον ε, Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και αν δεν κατάφερα να απαντήσω σε όλα σας τα ερωτήματα, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φαμπάλεκο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αυτή η πρώτη μας συνάντηση. Μας παρουσιάσετε τις δυνατότητες της ΕΤΕ στον γεωργικό τομέα. Καλή συνεννόηση με τον Επίτροπο Χόγκαν για τον γαλακτοκομικό τομέα, αλλά και για τους υπόλοιπους τομείς της γεωργίας. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας και τη διαθεσιμότητά σας για ε, μελλοντικές συναντήσεις. Όπως ξέρετε και σας είπε ο Πρόεδρος, εγκρίναμε τις συστάσεις των συντονιστών. Να σας υπενθυμίσω μόνο την επόμενη μας συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρίου το απόγευμα και την 1η Δεκεμβρίου πρωί και απόγευμα. Αυτά και λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας μεσημέρι.